Ε, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Πολλά υπάρχουν ε, στην Μεσιά Διάταξη και στις 10 ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων ε, θα έλθει εδώ και 9 με 10 δύο σημεία να εξετάσουμε ουσιαστικά τα, τι έχουν γίνει μέχρι, τι έχει γίνει μέχρι τώρα και μπορούμε να επανέλθουμε στο τέλος του πρωινού στην αποστολή μας, στην ταξίδι μας στην Ουγκάντα γιατί η UTM Σομελία και ο κ. Γκαλερ θα πριν από τις 10 το πρωί θα μας πει την κ. Σανκή στην απόψη ε, σχετικά με τις ε, κύριες προκλήσεις ε, και ε, θα ήθελα να σας κάνω ορισμένες ανακοινώσεις για τις επόμενες συναντήσεις μας. Την Πέμπτη το πρωί θα έλθει ο Βέλγος Υπουργός Άμυνος κ. Ντεκρέμ από την ε, Κατρίν Άστον έλαβε εντολή για να μας πει πώς έχει η κατάσταση στο Συμβούλιο, τι έγινε στο Συμβούλιο στην, με τους Υπουργούς Εξωτερικών και τους Υπουργούς Άμυνας. Ο κ. Ντεκρέμ λοιπόν θα έλθει εδώ και θα μας πει τι ακριβώς έγινε και η κυρία Γιανέλα ε, διευθύντρια για το USA η οποία θα έλθει επίσης και θα μας μιλήσει για τη Βόρεια Κορέα και το Ιράν και κλεισμένο το θηρόν συνάντηση με την αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν και τη χερσόνησο της Κορέας. Αύριο το πρωί θα έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων με, τον, με την Επίτροπο Τζόρτζεβα και θα ήθελα να σας πω πώς έχουν τα πράγματα με την αποστολή μας ε, το μήνα που μας πέρασε στο UATM Σομαλία και ταξίδι ήταν στην Ουγγάντα με τον Τζεμ Βαν Όρντεν, Ντεγιον Πάσκου και ο κ. Λουάν και εγώ συμμετείχαμε και στην αποστολή αυτή, στο ταξίδι αυτό επισκεφθήκαμε στο Μπιάνγκα στο στρατόπεδο αυτό που γίνεται η εκπαίδευση των ε, στρατιωτών της Σομαλίας και ε, με τη βοήθεια της ε, του στρατού της Ουγγάντα και δική μας και μετά συναντηθήκαμε στην Καμπάλα στο Γενικό Αρχηγείο και με πολίτες και στρατιωτικούς ε, και πέρασε καρπούς νομίζω, σύντομη συνάντηση αλλά ιδιαίτερα πυκνή και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επίσης ε, γιατί ήταν ας την αποκαλέσουμε μια ελαφρά αποστολή με 140 στρατιωτικούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά χαμηλό το κόστος, ε, αλλά που επηρεάζει ιδιαίτερα την κατάσταση και όσον αφορά την εκπαίδευση των στρατιωτών των Σομαλών. Επίσης πολιτικά επηρεάζει τα πράγματα στους εταίρους μας στην περιοχή, στην Ουγγάντα βέβαια, ξεκινώντα ε, πρώτα απ' όλα από αυτούς και οι αρχές οι δικές τους εξέφραν την ικανοποίησή τους που είμαστε εμείς εκεί και πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στη UTM και στη στρατό τη Ουγγάντα αλλά και όλοι οι άλλοι εταίροι οι οποίοι συμμετέχουν εκεί σε αυτή την ευαίσθητη περιοχή του κέρας της Αφρικής και οι Ηνωμένε Πολιτείε βέβαια που συμμετέχουν στην όλη διαδικασία και οργανωτικά, οικονομικά, η Αφρικανική Ένωση που με τη Μισόμ η οποία είναι εκεί στη Σομαλία, είναι στην πρώτη γραμμή του μετόπου, ας το πούμε έτσι, και επίσης Αιθιοπία, Κένια, Τζιμπουτί, αυτές οι χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια για τη σταθεροποίηση στη Σομαλία και μέσω αυτής της αποστολής εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχουμε σε αυτή την προσπάθεια την πολύπλευρη γενικότερα και πρόκειται για ένα σημαντικό πολιτικό κεκτημένο το οποίο θα πρέπει να εξακολουθήσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε και επίσης πέρα από την ιδιαίτερο επαγγελματικό χαρακτήρα, μπορώ να το πω αυτό εκ μέρους των συναδέλφων και των ε, στρατιωτών των Ευρωπαίων στην Ουγγάντα, να προσθέσω επίσης ότι παρατηρήσαμε και ορισμένες μικροβελτιώσεις που θα μπορούσαμε να επιφέρουμε πρώτα απ' όλα για τους ομολούς στρατιώτε ότι εκπαιδεύονται εκεί και από ό,τι μας είπαν οι στρατηγικοί της Ουγγάντα που είναι στην πρώτη γραμμή στη Σομαλία ε, σήμερα οι δυνάμεις Σομαλίας ε, οι ικανότητες τους ε, δεν είναι τόσο, η αποστολή τους δεν είναι τόσο στρατιωτική, στρατιωτικές οι αποστολές, αλλά οργανωτικές. Άρα λοιπόν μια εξέλιξη της όλης αποστολής και να εκπαιδεύουμε ε, και αξιωματικού για να πλαισιώνουν το στρατό. Αυτό είναι κάτι το θετικό και ορισμένοι από εμά επίσης ε, εξέφρασαν την έκπληξή τους ε, και εκδήλωσαν και τον ενδιαφέρον τους ε, για αυτή τη σειρά που φτάνει από ε, το πώς ε, έχουμε τους στρατιώτες αυτού μέχρι την ένταξή τους εκεί και ασχολούνται με την εκπαίδευση χωρίς να έχουν όμως λόγο στην επιλογή ούτε και στην επανένταξη επιλογή επανένταξη τι σημαίνουν ε, από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια κάποια παρουσία επιτόπου στη Σομαλία που από πολιτική πλευρά όμω δημιουργεί δυσκολίε σε αρκετά κράτη-μέλη. Και εμείς ε, θεωρούμε ότι κρίμα που η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αυτό το σημαντικό τομέα της εκπαίδευσης δεν έχει τίποτα να πει στο ξεκίνημα, στην επιλογή και στο τέλος στην επανένταξη αυτού του προσωπικού από τη Σομαλία και διαπιστώσαμε κυρίως ότι σε αυτό το τελευταίο, ε, στους τελευταίους στρατιώτες ε, τουλάχιστον 100 ε, στάλθηκαν στη Σομαλία μετά από ιατρικές εξετάσεις που απέδειξαν ότι ήταν κατάλληλοι ικανοί να υποστούν την εκπαίδευση που τους προτινόταν. Βέβαια η εκτίμηση αυτή, αυτόν το είχαν δει από την αρχή, τότε θα είχαμε γλιτώσει από παρόμοια πράγματα, γιατί καταλαβαίνετε ότι από οργανικής πλευράς υπάρχουν δυσκολίε να ε, διώχνει κανείς κόσμο στη συνέχεια. Αυτά λοιπόν, αυτές είναι οι απόψεις μας και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν και πολιτικές πιέσεις ε, που παίζουν το ρόλο τους ε, στην όλη αλυσίδα. Να δώσουμε το λόγο συναδέλφο που θα να βάλουν λόγο και η γραμματεία της Επιτροπή συνέταξε μια έκθεση, την έχετε την έκθεση και εγώ ίδιος θεωρώ ότι η αποστολή αυτή ήταν, στέφτηκε με επιτυχία και με έκανε, μου έκανε έκπληξη ε, ο λόγος κόστους αποτελεσματικότητας ε, γιατί με χαμηλά, με λίγα έξοδα Έχουμε εκεί αυτόν τον κόσμο που μας επιτρέπει να είμαστε σε σημαντική περιοχή, σε αυτή τη διαδικασία που αφορά τη Σομαλία. Γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει αναλάβει ρόλο ε, όσον αφορά ε, την πειρατεία στην περιοχή, μαζί με τους Αμερικανούς, την Αφρικανική Ένωση, με τον ΟΗΕ και τα κράτη του κέρατος Αφρικής, πρόκειται για μια προσθέμενη αξία πολιτική ιδιαίτερα σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ, ίσω ορισμένοι οι συνάδελφοι θέλουν να είναι περισσότερο επιβλακτικοί, Πάντω, ε, έχω θετική άποψη για να συνεχιστεί αυτή η αποστολή με τι βελτιώσεις βέβαια αυτέ που είπαμε και να δούμε αυτή την εκπαίδευση και για τους εξωματικούς ε, της Σομαλίας που πλαισιώνουν τους στρατιώτες. Να τονίσω επίσης ε, σαφέστατα το ενδιαφέρον των ε, αρχών της Ουγκάντα και στρατιωτικών και πολιτών. Μας έκανε πολύ καλή ε, ε, εντύπωση και το Γενικό Επιτελείο της Ουγκάντα ήταν παρόν για να σας δείξουμε πόσο συμμετέχουν οι Ουγκαντέζοι και πολύ σωστά θα ήθελαν να πλαισιωθούν, να υποστηριχθούν σε αυτή την προσπάθειά τους και από άλλες επίσης αφρικανικές χώρες που έδωσαν ε, δικά του ε, στρατό, προσέφεραν στρατιωτικά τμήματα επίση, αυτό και είναι και στην πρώτη γραμμή στο μέτωπο της Ομαλία, Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι υποστήριξη θα μπορούσε να δοθεί στην Ουγγάντα. Αυτά θα ήθελα από δική μου πλευρά να σα πω. Ο κ. Βανόρντεν ε, που ήταν και εκείνο παρόν στην αποστολή αυτή θα ήθελα να σα πει μερικά πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως ήταν μια εξαιρετικά καλά οργανωμένη επίσκεψη και πολύ ευχάριστη. Το βασικό ήταν το θέμα της ε, ισχύουσας ε, κατάστασης στην ε, Καμπάλα που διαπιστώσαμε αφού φτάσαμε και βλέπουμε ότι τώρα η ε, Ουγγάντα είναι στις ε, επικεφαλίδες των εφημερίδων. Ε, βέβαια είδαμε ιδίω τρία ουσιαστικά θέματα που πρέπει να διερευνήσουμε. Το ένα είναι η απόδοση των στρατιωτικών δυνάμεών μας, διότι ε, δεν ε, είδα κανέναν ε, κοινοτικό στρατιωτικό, είδα Ισπανούς, είδα από άλλες χώρες και ε, αν κρίνουμε το τι κάνουν καλό θα ήταν να τους πούμε ότι εφόσον μιλάμε ε, για τους ε, επαγγελματίες εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ε, να πηγαίνουν τα πράγματα πολύ καλά στην Ουγγάντα και άρα δεν εξεπλάγει όταν είδα ότι ε, εργάζονται σωστά. Βεβαίως υπάρχει καλή συνεργασία με την ε, Ουγγάντα και όντως ε, έχουμε άτομα τα οποία αναχωρούν από τη Σομαλία και με το αλεξίπτωτο καταλήγουν στην Ουγγάντα ε, για να καταλάβετε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει. Υπάρχει προσπάθεια να έχουμε μη επαγγελματίες αξιωματικούς και από εκεί να επιλέξουμε από τους οκάντα ορισμένους αξιωματικούς πράγμα το οποίο δεν είναι πολύ εδαφικό και αυτό είναι που προσπαθήσαμε να κάνουμε Οπότε το πρώτο είναι η επίδοση της Επιτροπής και βεβαίως το δεύτερο βασικό είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αυτής καθιαυτής διότι από ό,τι αντιλαμβάνομαι αυτή ήταν μια επιχείρηση η οποία καταρχήν έπρεπε να ε, είναι μια επιχείρηση εκπαιδευτική που θα ξεκινούσε από το Τζιμπουτί, κατέληξε στην Ουγκάντα. Ε, η ε, Ουγκάντα είναι ευτυχής που βρισκόμαστε εκεί, αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά ειδικά να βρίσκεται εκεί διότι οι νεοσύλλεκτοι ε, επιλέγονται και πληρώνονται από τις Ηνωμένε Πολιτείες και υπάρχει και ε, στήριξη στρατιωτικής μέρημνας και διοικητικής μέρημνας από τις Ηνωμένε Πολιτείε και το πνεύμα της εκπαιδεύσεως διέπεται από τη φιλοσοφία των Ηνωμένων Πολιτειών με τις οποίες υπάρχουν και άλλες συνεργασίες. ένα λόγο γιατί πρέπει να είμαστε εκεί. Αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχει μία πιο συλλογική ε, αντιμετώπιση, δηλαδή ε, σαν να έχει ορισμένα ε, ε, ε, δικαιώματα στον όρο αυτό ο η Ευρωπαϊκή Ένωση να τον έχει επινοήσει αλλά υπάρχει εδώ και μερικές δεκαετίες ε, ένα ερωτηματικό στο τι σημαίνει comprehensive approach, μια συλλογική προσέγγιση διότι η αντιπροσωπεία στην Καμπάλα ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχει ούτε καν επισκεφθεί ε, εις την στρατιωτική αποστολή. Αυτό όσον αφορά την comprehensive approach, δηλαδή τη συλλογική αντιμετώπιση όπως την αντιλαμβάνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε δεν βλέπω κανένα λόγο γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτή την αποστολή. Ε, το επόμενο είναι περί τίνος ομιλούμε και υπάρχει συνεργασία και στη Σομαλία. Δεν πήγαμε μεν στη Σομαλία και βασιζόμαστε σε άλλους για να μας πούν ε, τι συμβαίνει στη χώρα αυτή, αλλά αυτό που μας ελέγχθη σαφώς και ε, από κατοίκους της ε, Ουγκάντα είναι ότι η αποστολή στην Ουγκάντα δεν είναι επαρκής διότι η εντολή του ΟΗΕ ήταν για 12 άτομα οι οποία ποτέ δεν επετεύχθη. Στην Ουγκάντα μας λέγουν ότι χρειάζονται 20.000 για να γίνει σωστά η δουλειά. Οπότε υπάρχει μία ανεπαρκής ε, αποστολή της, της, των Ηνωμένων Εθνών. Υπάρχει και αποστολή... Ε, των Αφρικανικών κρατών από τον Μπουρούντι και την ε, Ουγγάντα και το θέμα είναι πόσο θα αμυφθούν αυτοί οι στρατιώτες ορισμένοι ε, πληρώνονται με αμερικανικούς μισθούς πράγμα το οποίο είναι μια πολύ δαπανηρή άσκηση. Όσον αφορά την κατάσταση που διαπιστώσαμε και τα τεκτενόμενα στο Μαγαντίσου δεν ξέρουμε ακριβώς τι συμβαίνει αλλά προηγούμενες αποστολές περιελάμβαναν ε, πολλούς ε, λιποτάκτες και πολλούς απόντες ε, οι οποίοι εξαφανιζόντουσαν διότι νομίζω έμεναν απλήρωτοι κάθε εβδομάδα ενώ τώρα υπάρχει ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος αμοιβή αυτών των στρατιωτών και άρα περισσότερες πιθανότητες να παραμείνουν αλλά δεν ξέρουμε πόσο αποτελεσματικοί είναι πότε θα ξαναγυρίσουν στο Μογκαντήσου, αν έχουν ενταχθεί σε άλλες μονάδες που είναι ήδη εκεί ή εάν έχουν δημιουργήσει αυτοτελείς μονάδες, τίποτα από όλα αυτά δεν είναι πολύ σαφές. Αυτό που αντιλαμβάνουμε όμως είναι ότι η αν εχουν δημιουργησει αυτοτελεις μοναδες τιποτα απο ολα αυτα δεν ειναι πολυ σαφες αυτο που αντιλαμβανουμε ομως ειναι οτι η κατασταση στο Μογκαντήσου είναι πάρα πολύ σοβαρή και υπάρχει και στενή σχέση με την πειρατεία η οποία ε, διεξάγεται εκεί. Αυτό διεφάνει. Άρα η ε, επίσκεψη ήταν πολύ χρήσιμη, πολύ αποτελεσματική, πολύ καλά οργανωμένη. Ε, συγχαίρω τους στρατιωτικούς οι οποίοι ε, έχουν αναπτυχθεί εκεί που είναι υπό την ηγεσία των Ισπανών, συνεργάζονται καλά. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μία, ένα πραγματικό ρόλο και νομίζω ότι η η επιχείρηση στη Σομαλία είναι διαφορετική και θέτει πολλά ερωτηματικά που μας ανησυχούν. Μάλιστα. Το θαύμα της πολιτικής είναι όταν από την ίδια διαπίστευση για το πόσο εξαιρετική ήταν αυτή η αποστολή καταφέρνουμε να καταλήξουμε σε εντελώ διαφορετικά αντίθετα αποτελέσματα για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι να σας πω, εγώ το βρίσκω αυτό πολύ τιμό και δεν μπορώ να καταλάβω τι θα έκανε το ΝΑΤΟ στην Ουγγάντα. Είναι στο Αφγανιστάν, είναι, στη, είναι στο, στη Λιβύη και έχει πάρα πολλά πράγματα να κάνει. Είδα 40.000 ε, ε, στρατιωτικούς ε, στην, στην περιοχή και μάλιστα είδα και το, το, το σήμα τους, το φορούσαν, το σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μα αυτό είναι το μόνιμό μου πρόβλημα ότι μόνο σε αυτό, σε ένα μπλε στίκερ ουσιαστικά περιορίζεται το, ε, η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ουσιαστικό ως ε, εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Μάλιστα, λέει ο κύριος Ντονζό. Συμφωνώ στην παρακολούθηση των ε, κληρωτών και στην επανέντοξη, στην επανέντοξη, στην επανέντοξη τους. Είναι γεγονός ότι δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε ως προς αυτό, δημιουργεί πρόβλημα η στάση αυτή και νομίζω ότι και οι πράσινοι συναδελφοί μας μας είχαν θέσει πολλές φορές σε αυτό το θέμα της επιλογής των κληρωτών και την ενδεχόμενη ε, μάλιστα στράτευση κληρωτών ε, κάτω από την, την ηλικία της ενηλικίωσης, κάτω των 18. Είναι ένα πρόβλημα και όταν υπήρχε αυτή η περίπτωση, ε, όταν ήταν ανήλικη δηλαδή η κληρωτή ή που η ιατρικής απόψεως ε, δεν ήταν επαρκής, ε, ίσω θα έπρεπε να μην επιλέγονται. Ήταν ένα από τα σημαντικά ζητήματα, ένα από τι σημαντικέ προκλήσεις και είχαν αναφερθεί πολλές φορές στην συγκεκριμένη Επιτροπή. Ο κύριος Φάγκελ θέλει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να θέσω ορισμένα ερωτήματα, ορισμένα ζητήματα, τα οποία βέβαια έθεσε ήδη ο κύριος Φανόρντεν. Εγώ Χαίρομαι με τον τρόπο με τον οποίο έθεσε ορισμένους προβληματισμούς για την ε, εμπλοκή μας. Θα ήθελα καταρχάς να σας επενέσω για την οργάνωση της αποστολής αυτής. Ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ, ε, πολύ περιεκτική και η σύνοψή σας, η επισκόπησή σας είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης να ενημερωνόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε συνεχώς για αυτές τις μακρινές αποστολές τις οποίες ε, ε, έχουμε ξεκινήσει να μην τις εγκαταλείπουμε δηλαδή. Κάτι τέτοιο βέβαια σημαίνει σταθερή πολιτική δέσμευση και υποστήριξη και ακόμη Και αν δεν χρειάζεται πια να είμαστε παρόντες κάπου, χρειάζεται και μία απόφαση για να αποσυρθούμε. Δεν έχουμε φτάσει βέβαια ακόμη σε αυτό το επίπεδο σύμφωνα με όσα είπατε εσείς και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας. Ήταν μία μάλλον ε, ε, εμπνευστική αποστολή και συνεπώς πολλά πράγματα μπορούν να προκύψουν από αυτήν. Ένα θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι το πρόβλημα της πειρατείας και τον, ε, το θέμα της ε, κοινωνικής και οικονομικής αιτίας ε, αυτού του προβλήματος. γιατί ένα μεγάλο τμήμα του ε, λαού της ε, Σομαλίας ε, βγάζει το ψωμί του έτσι και δεν θα έπρεπε να είμαστε επικεντρωμένοι τόσο πολύ. με το να βλέπουμε ποιο είναι το πρόβλημα που δημιουργείται στο διεθνές εμπόριο, αλλά θα έπρεπε να μας απασχολεί και ιδιαίτερα για ποιο λόγο υπάρχει αυτό το πρόβλημα και επίσης πού πηγαίνουν τα κέρδη της πειρατείας και κατά πόσο βέβαια αλλάζουν τα πράγματα στο σύνολο της Αφρικανικής Υπήρου λόγω της παρουσίας μας ε, με διάφορους τρόπους και μέσω διαφόρων αποστολών. Επίσης, κάθε φορά που πηγαίνουμε να εξετάσουμε πώς, πηγαίνουν τα πράγματα ε, με τις δικές μας αποστολές, τις αποστολές των Ηνωμένων Πολιτειών ή διάφορες, διάφορα άλλα ζητήματα, ε, ίσως θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες της Αφρικανικής Ένωσης ε, να αναλάβει και εκείνη το μερίδιο της ευθύνης της. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε λοιπόν μια εκτενή συζήτηση με την Αφρικανική Ένωση ε, στο μέλλον για τη στρατηγική, την αναπτυξιακή στρατηγική, τη στρατιωτική στρατηγική, τα ζητήματα ασφαλείας, γιατί θα έπρεπε να είναι ένας βασικός παίκτη στην περιοχή και θα έπρεπε να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη. Οπότε, να σας ευχαριστήσω και πάλι για την έκθεσή σας, αλλά και για την αποστολή και πιστεύω ότι θα έπρεπε να συνεχίσουμε να είμαστε ε, παρόντες ε, στην ε, συγκεκριμένη περιοχή. Εντάξει, για την Αφρικανική Ένωση, να πούμε για το σημείο αυτό, ναι, προετοιμάζουμε μια συζήτηση για αυτό το θέμα, της 30 Ιουνίου και θα έχουμε αρκετούς προσκεκλημένους ε, για να μπορούμε ακριβώς να δούμε τις εταίρους μας ε, στο στρατιωτική πτυχή και αυτό μας το υπενθύμησαν και οι στρατιωτικές αρχές της Ουγκάντα ότι η ανάμειξη στη Σομαλία είναι και καθοριστική αλλά και κενά και βασίζεται σε δύο αφρικανικά κράτη αυτή τη στιγμή που ζητούν ε, την υποστήριξη και των υπόλοιπων κρατών ε, που θέλουν να βοηθήσουν. Ε, είναι μια σημαντική συζήτηση που προσπαθούμε να οργανώσουμε τις 30 Ιουνίου. Ο κύριος Πασκού, μέλος επίσης της αποστολής της αντιπροσωπείας αυτής και μετά πάμε στο επόμενο σημείο γιατί πριν από τις 10 θα πρέπει να το εξετάσουμε. Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι συμφωνώ απολύτως με το αποτέλεσμα της έκθεσης, δηλαδή ότι είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη ε, επιχείρηση η οποία δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρή και η οποία είναι πολύ απαραίτητη. Από ό,τι κατάλαβα έχουν γίνει οι απαραίτητες, οι απαραίτητοι διακανονισμού. Εγώ προσωπικά ε, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά για ποιο λόγο όταν δεν συμμετέχει η Ευρωπαϊκή, Ευρωπαϊκή Ένωση ε, την κατακρίνουμε που δεν συμμετέχει και όταν συμμετέχει λέμε ή ότι δεν είναι επαρκής η συμμετοχή ε, ή ότι δεν είναι ε, ρόλος της. Ίσως θα έπρεπε πιστεύω να ε, είμαστε λίγο πιο ρεαλιστές να αξιολογούμε την κατάσταση και να προσπαθούμε να δούμε, να δούμε την αξία και για την κατάσταση στην περιοχή, αλλά και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν βέβαια και άλλες ε, πτυχές ε, της ε, ΚΕΠΑ που χρήζουν συζητήσεως, αλλά κατά την άποψή μου νομίζω ότι η σχέση αποτελέσματος και κόστους είναι μεγάλη. Εντάξει, παρακαλώ τον Βαμόρνταν και τον Ζαμπασκού, οι οποίοι και συμμετείχαν ιδιαίτερα ενεργά, ε, έδειξαν την πείρα που διαθέτουν πάνω σε αυτό και ήταν κάτι το πολύ ευχάριστο. Και θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται με το επίπεδο εμπειρογνωμοσύνη της συγκεκριμένης αποστολή Νομίζω ότι είχαμε μία επιτόπου επίσκεψη υψηλή ποιότητας και γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες και να ευχαριστήσω και τους δύο ε, παρόντες σήμερα συναδέλφου ε, που είχαν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιτυχή έκφαση της αποστολή και επιμένω λοιπόν ότι ήταν μια πολύ εστιασμένη ε, επίσκεψη με πολύ ε, υψηλό βαθμό εμπειρογνωμοσύνη. Περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης πριν από τη συζήτηση με τον κύριο Βεστεβέλε που αφορά ε, την ε, γνωμοδότηση για την αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η κυρία Χάνκης, η οποία είναι αρμόδια για την Επιτροπή μας ε, ε, για την σύνταξη της γνωμοδότησης αυτής, όμως δεν είναι εδώ σήμερα, οπότε ο κύριος Γκάλερ θα την, θα την αντικαταστήσει. Μήπως μπορείς λοιπόν, Μίκαλη, να μας πεις σε γενικές γραμμές τα σημεία της έκθεσης αυτής, γιατί σήμερα το απόγευμα θα ψηφιστεί στην ΑΦΕΤ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αρνό και συγγνώμη που άργησα, δυστυχώς άργησε το αεροπλάνο από το Βερολίνο και συγγνώμη αν χρειάστηκε να αλλάξετε λίγο την ημερήσια διάταξη. Πράγματι δεν είναι εδώ η κυρία Χάνκης και μου ζήτησε να σας παρουσιάσω την γνωμοδότησή της. Η γνωμοδότηση επί του σημείου αυτού έχει συνταχθεί από και από οπτικής γωνίας ε, ε, και πα και αφορά τα εξωτερικά στοιχεία της αντιτρομοκρατικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η συγγήτρια. θέλει να τονίσει ειδικότερα τη σημασία της πολιτικής αυτής, τη σημασία του ρόλου της ευρωπαϊκής στρατηγικής, όπως επίσης αλλά και της, της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας και τη εναρμόνισης των δύο, δύο, δύο αυτών στοιχείων. Διατλαντική σχέση, αναφορά σε συγκεκριμένες περιοχές και αναφορά στο γεγονός ότι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για την αντιμετώπιση των τραμοκρατικών ε, δραστηριοτήτων, όπως επίσης και το γενικό πλαίσιο που θέτουν ε, τα Ηνωμένα Έθνη. Τονίζει επίση ε, την σημασία συντονισμού και συνεργασίας με τον ΝΑΤΟ, αναφέρεται στη σχέση του Διεθνούς Οργανωσμένου Εγκλήματος της Λαθρεμπορίας Ναρκωτικών ε, όπως επίσης και της τρομοκρατίας και τονίζει τον ε, απαραίτητο ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετω... τον απαραίτητο ρόλο του ε, συντονιστή αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστεί τους συναδέλφους για τις ε, τροπολογίες της. Έχει προσπαθήσει να τις ε, συμπεριλάβει σε πέντε συμβιβαστικές τροπολογίες, ε, τις οποίες προτείνει να ψηφιστούν. Υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες οι οποίες προσπαθούν ε, δημιουργικά να επεκτείνουν ε, το πεδίο εφαρμογής συγκεκριμένης γνωμοδότησης μόνο εμέσως όμως ε, ή σε ζητήματα που αφορούν την εξωτερική διάσταση της αντιτρομοκρατικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης αναφέρει ότι δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι ο βασικός στόχος πολιτικής αυτής είναι να σώζει τις ζωές αθώων ανθρώπων. Δεν μπορούμε πάντοτε να αμβλύνουμε τις ε, ε, ε, βασικές, τις ριζικές αιτίες της αντιτρομοκρατικής τρομοκρατικής δράσης. Σε σχέση με τις τροπολογίες 6 της Βαρόνης Λάτφορντ και της 39 από την κυρία Γετεμέκη, προτείνει, προτείνουν ένα πάνελ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων για την αναθεώρηση των πολιτικών και το αναφέρει μάλιστα και η έκθεση της κυρίας Ίνετφελτ που είναι άλλωστε και ε, η ε, συντάκτρια της έκθεσης καθήλυν ε, αρμόδιας επιτροπής. Ρωτά λοιπόν η κυρία Χάνκης πώς θα είναι ανεξάρτητο αυτό το πάνελ, ποια θα είναι η μέθοδος του διορισμού των μελών του και ποια θα είναι τα κριτήρια για να δεχθούμε ή να απορρίψουμε έναν ε, τέτοιου είδους διορισμό, έναν διορισμό σε αυτό το πάνελ. Οπότε λοιπόν ε, ζητά να μην ε, υποστηριχθεί το σημείο αυτό. Επίσης, στο φάκελό σας θα δείτε και το κείμενο των πέντε συμβιβαστικών τροπολογιών Αυτό έχω λοιπόν να προτείνω εκ μέρου τη κυρίας Χάνκη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριο, κύριος Πασκού, επιθυμεί το λόγο. Πάρα πολύ σύντομα. Μου ζήτησε η ομάδα μου να πάρω το λόγο εκ μέρου τη ομάδας για να υποστηρίξω τις συμβιβαστικές τροπολογίες που παρουσιάστηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, κύριε Λούζιν. <coughs> Um, ευχαριστώ. Ήδη σε προηγούμενες συζητήσεις είχα αναφέρει ότι λυπάμαι πάρα πολύ ε, που δεν ε, έχουμε θεωρήσει ότι η αντιτρομοκρατική πολιτική που μας απασχολεί τόσο πολύ ε, δεν περι, γράφεται στη, στα αντιτρομοκρατικά θέματα και θα ήθελα να ληφθούν υπόψη τα σχόλια αυτά ή στις τροπολογίες που θα γίνουν. Επίσης διαπιστώνω ότι υπάρχει μία πληθώρα τροπολογιών οι οποίες είναι κριτικές έναντι των ε, μέτρων αντιτρομοκρατίας που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής, ιδίως όσο αναφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά και όσον αφορά την ε, ε, δύναμη η οποία ε, χρησιμοποιείται και ελπίζω ότι και αυτά θα περιληφθούν στην γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος θα επιθυμούσε το λόγο για το σημείο αυτό. Ίσως ο Μίκαελ, έτσι καταληκτικά. Ευχαριστώ για τη στήριξη την οποία ε, ανέφερε ο συνάδελφος Πάσκου εν ονόματι της πολιτικής του ομάδος. Νομίζω ότι όσον αφορά τη δεύτερη τροπολογία συμβιβαστικά έχουμε αναφέρει ότι ε, θα πρέπει κανείς ε, να καταπολεμήσει τις αιτίες. Αν όμως εδώ αναφερθούμε εις, ε, στις ε, συγκεκριμένες πτυχές αυτής της πολιτικής και τα μέτρα τα οποία μπορούμε να λάβουμε δεν είναι εδώ το κατάλληλο σημείο όπως άλλωστε ελέγχθη ε, για να γίνει μία λεπτομερής ε, μελέτη διότι ε, πρέπει να υπάρχει μια αντιτρομοκρατική πολιτική όπως λέγεται και εάν ε, λάβουμε μία σαφή θέση, τότε αυτό σημαίνει ότι όλες οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στην περιοχή από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνουν προληπτικά μια καταπολέμηση της τρομοκρατίας για να αποφύγουμε να οδηγηθούμε σε μια τέτοια κατάσταση και πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ βασικό άπτεται το θέμα αυτό και άλλων πολιτικών αλλά το πρόβλημά μας δεν είναι να επιλύσουμε όλα τα θέματα όλων των πολιτικών εδώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ε, να σα υπενθυμίσω κάτι μετά από τη συζήτηση αυτή που κάτι 11 θα ολοκληρωθεί μαζί με το ΕΦΕΤ. Σε... Θα έχουμε τον κύριο Ντεκερκόφ ε, συντονιστή για τη δημοκρατική δράση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα εξετάσουμε το θέμα μαζί του. Για 10 λεπτά θα διακόψουμε για να δούμε την επόμενη συνάντησή μας με την αφέντα ακριβώ. Γεια σας, μάλλον διάλειμμα για 10 λεπτά. Ε, Αγαπητοί συνάδελφοι, να καλωσορίσω τον Υπουργό Γκουίντο Βέστερβέλε. Χαρά μας να τον έχουμε εδώ. Θα είναι σίγουρα σημαντική αυτή η συνάντηση και τον συνάλφο πρόεδρο Ντανζό να ευχαριστήσω ο οποίος ε, γενναιόδωρα μας παραχώρησε χρόνο από την υποεπιτροπή του για να συναντηθούμε και να ακούσουμε τον Υπουργό. Σίγουρα είναι τη στιγμή που πρέπει αυτή η συνάντηση μαζί σας με την πρόσφατη υιοθέτηση από την Επιτροπή μας μια σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών για την προσεχή Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Μετά από λίγες μέρες από την οθέτηση από πλευρά της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ενός ψηφίσματος για τον ειδικό χαρακτήρα που αποδίδεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τα Ηνωμένα Έθνη γιατί ακριβώς εκπροσωπούν τα κράτη-μέλη σε θέματα κοινή εξωτερικής πολιτικής. Πρόκειται για επιτυχία της ευρωπαϊκής διπλωματίας που θα πρέπει σίγουρα να της αποδώσουμε την αξία που πρέπει. Και εδώ τοποθετείται η συναντήσή σας, σε, η επισκεψή σας σε ένα ένα πλαίσιο ευαίσθητο όπως το Μαγκρέμπ και στο Μασρίκ και το τι συμβαίνει τώρα στις αραβικές χώρες. Και καλούμεθα να δώσουμε μια κοινή απάντηση εκτός από απαντήσεις σύμφωνα με τις διμερείς μας σχέσεις. Κύριε Υπουργέ, ακριβώς συνάντησή μας σήμερα έχουμε να κάνουμε με στόχους και με την πείρα που διαθέτει η Γερμανία σαν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η Γερμανία, η χώρα σας, όπως το είχε κάνει και η Ιταλία, καταβάλει προσπάθεια για να δώσει μια αξία ευρωπαϊκή στην έδρα στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ιδιαίτερα ε, υποστηρίζουμε αυτές τις πρωτοβουλίες, ε, ιδιαίτερα πεπισμένοι ότι έχουν αξία και θα θέλαμε να δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες ε, τι ακριβώς συμβαίνει και στη σύσταση της Επιτροπής μας, ε, την οποία αναφέρθηκα πριν, εκφράσαμε την απόψη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας με την, μεταρρύθμι, με την αλλαγή του θα πρέπει να δώσει, να προσφέρει μια μόνιμη έδρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένοντας την επίτευξη του στόχου αυτού θα πρέπει να ισχύσει ένα σύστημα εναλλαγής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις μη μόνιμες έδρες του Συμβουλίου ασφαλείας. Ε, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν διαθέτουμε και ιδιαίτερα πολύ χρόνο ε, ε, και επειδή ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τα θέματα αυτά οι συνάδελφοι, δίνω τον λόγο πρώτα στον πρόεδρο Ντόνζον. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, εξ ονόματος της Επιτροπής ασφάλεια και άμυνα του Κοινοβουλίου μας. Σας καλωσορίζω και θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος ε, γιατί ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα να σας ακούσουμε και να συζητήσετε με τους συναδέλφους μας και να σας πω ότι θα ήθελα βέβαια να σας ακούσω για το θέμα της Λιβύης, το οποίο ε, και χάραξε το πρώτο εξάμεινο εδώ και στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως επίσης και την κάποια απογοήτευση εδώ στο Κοινοβούλιο μας για τους περισσότερους από εμά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθ' αυτή δεν μπόρεσε να παίξει ένα σοβαρό σπουδαίο ο ρόλο σε αυτό το θέμα τη Λιβύης και όσον αφορά την ε, στρατιωτική συνιστόσα, αρκετοί εδώ είμαστε υπέρ μια κοινή ε, πολιτική ασφάλεια και άμυνα, φιλόδοξη όπω προβλέπεται από τι ειδικές τη Αβώνα και εδώ και αρκετού μήνε ε, τι βλέπουμε, μια, παρατηρείται μια κάποια επιβράδυνση έτσι να το πούμε και βιενικά σε αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό ενδιαφερόμαστε να σας ακούσουμε πώς αντιλαμβάνεστε αυτή την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και πέρα από το θέμα της Λισβής αρκετές πρωτοβουλίες που προσπαθούν να, όπως από πλάς Γερμανίας, Σουηδίας, το Μετσέριν, όλα αυτά και το τρίγωνο της Βαϊμάρης, Πολωνία, Γαλλία, Γερμανία. Θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεστε πάνω σε αυτό και αν ε, θεωρείτε ότι μπορούμε να ξαναξεκινήσουμε όπως πρέπει, γιατί η Γερμανία είναι και σημαντικός εταίρος, αλλά κάπως ε, έχει επιβραδύνει την δράση του. Εντάξει, εδώ λοιπόν και από πλευρά τη Επιτροπή μα και να λάβετε το λόγο ανάμεσά μα να χαιρετήσω για τη ζήτηση αυτή ε, ε, την παρουσία τη κυρία ε, από τη Βουλγαρία Υφυπουργό Αμήνα εδώ που ήταν στο συνέδριο συνάντηση Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνα και Ντάμιαν που είναι ο κόπτη Επίσκοπο τη Γερμανίας και που εκπροσωπεί τον αρχιεπίσκοπο της Γερμανίας. Ξέρουμε ότι η μειονότητα, η κοπτική ιδιαίτερα ενδιαφέρεται γι' αυτό και εκφράζει το ενδιαφέρον τη αυτή εδώ στην Επιτροπή μας. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις, διότι η ε, η Γερμανία θα αναλάβει την ε, πέμπτη συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφαλείας και αυτή η ε, θέση αναλαμβάνεται σε μια ταραγμένη εποχή σχετικά με τον αραβικό κόσμο, την Αφρική και έχουμε κοινά συμφέροντα η γυτνίασή μας αυτή να διεξάγεται δημοκρατικά και ειρηνικά. Πρέπει όμως να πούμε ότι αυτό το οποίο ξεκίνησε εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί. Ε, είμαστε στα πρώτα μέτρα μία πορεία στην οποία να διαπιστώνουμε αυτή τη στιγμή και βλέπουμε ότι ο προδιαγεγραμμένος δρόμος περιλαμβάνει όλο και περισσότερες διαμάχες και εδώ αναφέρομαι στη νότιο και στην περιοχή νοτιού και βορείου Σουδάν για να αναφέρω το πιο πρόσφατο παράδειγμα έχουμε άλλα θέματα τα οποία θεωρούμε παρελθόν αλλά ανέρχονται μόνο σε λίγες ε, ημέρες. Ε, η ε, Μέση Ανατολή, το Πακιστάν, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και της Βορείου Κορέας, η πειρατεία της της ακτές της Ανατολικής Αφρικής και ε, όλα αυτά ε, είναι θέματα που απασχολούν πολύ το Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά από ό,τι αντιλαμβανόμαστε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι κάτι παραπάνω από ένα, ένας οργανισμός διαχείρισης κρίσεων διότι πρέπει να προστατεύσει ε, την θέση του σε γενικότερα θέματα τα ανθρώπινα δικαιώματα, την εγκαθίδρυση της ε, ασφαλείας και της ειρήνης και γι' αυτό με το πνεύμα αυτό εμείς θα αναλάβουμε τη θέση μας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και με, αυτήν, ε, με αυτό το σκεπτικό θα αναλάβουμε την Προεδρία τον Ιούλιο για να διαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση διότι κατά τη γνώμη μας και ο ΙΕ πρέπει να ανανεωθεί και αυτό είναι ένα πολύ βασικό έργο το οποίο λοιπόν τώρα με την προεδρία του κυρίου Ντάις στην Ολομέλεια συζητείται, δηλαδή η μεταρρύθμιση του ΟΗΕ διότι ο ΙΕ και στο μέλλον θα πρέπει να έχει επαρκές κύρος και να είναι αποδεκτό σαν οργανισμός και αν δεν αντικατοπτρίζει την αρχιτεκτονική του σημερινού κόσμου άλλες μορφές όλο και περισσότερο θα αναλάβουν μέρος εκ των καθηκόντων του ΟΗΕ δηλαδή εδώ δεν πρόκειται για εθνικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να επιζητεί κανείς κατά την μεταρρύθμιση του ΟΗΕ αλλά ο οργανισμός αυτός να αντικατοπτρίζει καλύτερα την παγκόσμια κατάσταση από ό,τι μέχρι τούδε. Παραδείγματο χάρη, η Λατινική Αμερική δεν έχει μόνιμη εκπροσώπηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας όπως και η Αφρική και επίσης η Ασία εκπροσωπείται και όλα αυτά δείχνουν ότι η παγκόσμια τάξη εμφανίζεται περισσότερο έτσι όπως διαμορφώθηκε ε, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και γι' αυτό θα πρέπει να αναλυφθούν και άλλες ευθύνες από τον οργανισμό. Ε, υπάρχουν και άλλες προκλήσεις. Θα πρέπει ε, ο οργανισμός να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών όσον αφορά το δημόσιο δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, να μπορεί να προστατεύει του τους λαούς από τις παρεκτροπές ε, των κυβερνήσεων και αυτό είναι κάτι το οποίο διαπιστώνουμε. Η παγκοσμιοποίηση διαπιστώνεται και ε, αντικατοπτρίζεται αυτή την εποχή όχι μόνο σαν παγκοσμιοποίηση της οικονομίας αλλά και των αξιών, των απόψεων, του τρόπου ζωής αλλά και ιδίω αξιών. Και επειδή η Ευρώπη θεωρεί ότι είναι μία κοινότητα αξιών και ε, δικαιωμάτων ε, γι' αυτό και θέλουμε να αντιλαμβανόμαστε και τον ΟΗΕ μια τέτοια ενότητα ε, θα πρέπει επιπλέον να είμαστε έτοιμοι για το μέλλον διότι εμείς θέλουμε να υπάρχει πολυμορφία ε, και ε, έχουμε ζωτικό συμφέρον να προωθήσουμε την αρχή αυτή. Θα πρέπει να υπάρχει εκπροσώπηση της Ευρώπης και αναγνώρισή της από τα Ηνωμένα Έθνη και πρέπει να επισημάνουμε τις επιτυχίες. Το την, ε, ε, ε, την εξωτερική επιτροπή ε, υπηρεσία της Κάθρις Άσνον η οποία δεν έχει φτάσει ακόμη το επίπεδο το οποίο θέλουμε αλλά από πέρσι το Σεπτέμβριο πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει προοδοί οι οποίες πρέπει να διακηρύσσονται και ίσως η Ευρώπη δεν προβάλλει προς τα μέσα τις υπηρεσίες αυτές. Εγώ θεωρώ ότι η υπηρεσία αυτή είναι μία επιτυχία για την Ευρώπη και ε, θεσμικά μπορεί να αποδείξει ότι έχουν γίνει πρόοδοι έχουμε και ένα άλλο κοινό συμφέρον στην Ευρώπη πέραν της συνθήκης της Λισαβόνας αλλά πρέπει να έχουμε μία κοινή πολιτική ασφαλείας και ανέφερα και άλλες ε, επιτυχίες τις οποίες πρέπει να τονίσουμε τις διάφορες μορφές ε, αγαπητέ ε, συνάδελφε αναφερθήκατε σε, τρεις, σε τρία θέματα καταρχήν το το τρίγωνο της Βαϊμάρης ε, ο Πολωνικός Γερμανός, ο Πολωνός Γερμανός και Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών και την ε, προηγουμένη αυτή της συναντήσεως υπήρξαν ε, και άλλες συναντήσεις στο Καλίνιγκραντ μεταξύ του Πολωνού Υπουργού Εξωτερικού και μου από κοινού με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και νομίζω ότι συμφωνούμε και αυτή τη στιγμή ε, υπάρχει το ε, ε, επίκεντρο της προσοχής ή στη Μεσόγειο αλλά αν θέλουμε να έχουμε μία προοδευτική εξωτερική πολιτική δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ανατολικούς γειτόνους μας υπάρχει αυτή, αυτός ο θύλακος όπου συναντηθήκαμε με τον Ρώσο ομόλογό μας και η διαδικασία αυτή δεν έχει μόνο συμβολική σημασία αλλά αποτελεί όντως μία πρόοδο η οποία πρέπει να αναγνωριστεί. Ε, δεν συμφωνούμε σε όλα τα θέματα, δεν έχουμε επιτύχει όλους τους στόχους μας γιατί θα θέλαμε ε, να υπάρχει η αρχή της ευθύνης για ασφάλεια που να γίνει αποδεκτή από όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας Ξέρετε ότι στην τελευταία ψηφοφορία εμείς δηλώσαμε αποχή, είναι δύσκολο, αλλά εφόσον υπήρχε μία απόφαση για στρατιωτική εμπλοκή, εμείς ήμασταν της γνώμης ότι έπρεπε να αναλυφθούν πολιτικά μέτρα και είχαμε ε, καλούς λόγους να ακολουθήσουμε τη στάση αυτή, εξίσου καλούς λόγους με αυτούς τους οποίους πρόβαλαν άλλα μέρη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ε, θεωρώ ότι πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αισθάνεται μία διεθνή ευθύνη και βλέπετε ότι η χώρα μου δείχνει την στάση αυτή στο Αφγανιστάν και όχι μόνο πρέπει τώρα να επιζητήσουμε μια πολιτική λύση για την Λιβύη, να σταματήσει το καθεστώς του Καντάφη και να δημιουργηθεί χώρος για μια νέα αρχή. Αυτή η επιθυμία για νέα αρχή ε, συγκεντρώνει τις επιθυμίες πολλών λαών όπως και των αραβικών χωρών και μέση Φεβρουαρίου είχα συντάξει μία επιστολή επί του θέματος για την συνεργασία πληροφοριών ε, που υιοθετήθηκε από τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εξωτερικών και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα πέραν ε, της ε, πολιτικής συνεργασίας θα πρέπει να συνεργαστούμε με τις ε, δημοκρατικές χώρες πέραν της κοινωνίας των πολιτών και στα ιδρύματα όπως συζητήσαμε εχθές θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη πολυμορφία και ποικιλία και θα πρέπει να εξετάσουμε την δημοκρατία αραβική επανάσταση στην Τινησία ή στην Αίγυπτο και όχι μόνον, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται ακόμη στην αρχή, χρειάζονται πολύ δρόμο ακόμη και σαν Ευρωπαίοι δεν πρέπει να στηρίζουμε μόνο με καλά λόγια, αλλά είναι καθήκον μας να κάνουμε μία συγκεκριμένη προσφορά όσον αφορά την συμμετοχή στις αλλαγές μέσω του εμπορίου, μέσω επενδύσεων και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει συγχρόνως να ανοίξει τις εσωτερικές της αγορές για προϊόντα από τις χώρες αυτές που έχουν προσχωρήσει στη δημοκρατία κατά τρόπον ώστε να υπάρχει ένα μέρισμα που να προσφέρει η ελευθερία διότι στο τέλος έτσι μόνο θα μπορέσει να αποφασιστεί η βιωσιμότητα της διαδικασίας αυτής. Εάν δηλαδή η δημοκρατία μπορεί να επιτύχει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για αυτούς τους λαούς και ε, εφόσον ε, συζητήσαμε το θέμα αυτό δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για δημοκρατία αλλά και ε, για δυνατότητες καλύτερης διαβίωσης που αποτελούν ένα βασικό στοιχείο εις ε, την εξωτερική μας πολιτική και στις δυνατότητες ε, πολιτικής γυτνιάσεως. Όσον αφορά το Συμβούλιο Ασφαλείας θα ήθελα να σας πω ότι λαμβάνω υπόψη όλα αυτά τα θέματα και μέχρι τον Ιούλιο Πρέπει να σας πω ότι ε, θεωρούμε ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας δεν έχει δώσει τη δέουσα προσοχή στα θέματα αυτά μέχρι στιγμής και δεν χρειάζεται να σας πω πόσο σημαντικές είναι οι διαπιστώσεις αυτές για την Ευρώπη. Ε, ε, επιπλέον όμως για τον Ιούλιο θα πρέπει να προβλέψουμε όχι μόνο συζητήσεις για τις κλιματολογικές αλλαγές αλλά συγχρόνως και ε, για το δεύτερο θέμα, δηλαδή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κατά τη γνώμη μας αυτό δεν πρέπει να εξεταστεί μόνο σε σχέση με την Αραβική Άνοιξη και δεν αποτελεί ε, πρόκληση μόνο στον τομέα αυτό αλλά και στον γενικό τομέα της πολιτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζητήσαμε μία ενίσχυση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την ε, Ευρώπη, για τη σχετική στρατηγική διότι θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε παραδείγματο χάρη τα παιδιά στι ένοπλε σειράξει, και αυτό να επιτευχθεί μέσω της αναλήψεω ευθυνών μας στον τομέα αυτό. Δεν είναι μόνο μία επιταγή ε, που επιβάλλεται από τους συνανθρώπους μας αλλά για ένα επίγον θέμα και ε, ζητούμε να υπάρξει ένα ψήφισμα που να αναφέρεται εις ε, τις επιθέσεις σε νοσοκομεία που πρέπει να θεωρηθούν σαν βάρβαρες πράξεις. Ε, έχουμε όμως πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για να επιτύχουμε τους στόχους μας στον τομέα αυτό. Και τώρα φτάνω προς το τέλος μου και πρέπει να σας πω ότι επιπλέον θα ασχοληθούμε με πολλά επίκαιρα θέματα που είναι δύσκολα διότι υπάρχει η, τον Ιούλιο η πρόβλεψη της διακήρυξης ανεξαρτησίας του Νοτίου Σουδάν, κάτι που παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία και χθες ο Υπουργός Εξωτερικών ε, από κοινού, οι Υπουργοί Εξωτερικών αναφέρθηκαν ε, σαφώς επί του θέματος αυτού παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις εξελίξεις στο χώρο αυτό διότι πρέπει να αποφύγουμε μία κλιμάτωση της βίας στο χώρο και όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και ο ΙΕ ε, άμεσα πρέπει να τοποθετηθεί στο θέμα αυτό και να πιέσει κατά τρόπον ώστε να μπορέσει να ε, επιστρέψει ε, ο πληθυσμός της περιοχής αυτής στα σπίτια του και τέλος θέλω να σας ευχαριστήσω διότι έχω την εντύπωση ότι είναι απαραίτητο να ασχοληθούμε με τα θέματα τα οποία, ε, επί των οποίων δεν υπάρχει μία κοινή θέση αλλά ακόμη και εκεί που υπάρχει μία κοινή αντιμετώπιση στην Ευρώπη ε, θα πρέπει αυτή να παρουσιάζεται ως κοινή. Δηλαδή ε, ε έχουν αποφα... αποφασίστηκαν σημαντικές κυρώσεις για τέσσερα χρο τις χώρες, τη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράν και την Λευκορωσία και αυτό αποδεικνύει ότι ασχολούμεθα με τα ανθρώπινα δικαιώματα και αντιλαμβανόμαστε στην Ευρώπη ότι πρέπει να κινούμαστε ε, από κοινού και να αναλαμβάνουμε τις δεσμεύσεις μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και προσβλέπω στη συζήτηση που θα έχουμε. Θα ήθελαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Υπουργό. Συνάδελφοι, σύμφωνα με ότι, ότι συνηθίζεται θα έχουμε δύο γύρους παρεμβάσεων. Πρώτα οι συντονιστές και ο εισηγητής και ο πρόεδρος της ομάδας εργασίας για τις σχέσεις ανάμεσα στους δύο, ο συνάδελφος Σλάντορφ, Σλέντορφ. Και στον πρώτο αυτό γύρο θα έχουν από δύο λεπτά ο καθένας για να εκφραστούν. Ο πρώτος ομιλητής τον γνωρίζετε όλοι σας, είναι ο Χέρμαν Μπροκ. Έχει τον λόγο. Ο Μπροκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε σε αυτή την υποεπιτροπή δεν επρόκειτο να θεωρήσω ότι είμαι ένα συντονιστής και χαίρομαι κύριε Υπουργέ που είστε εδώ σήμερα και μιλήσατε για το ρόλο του Συμβουλίου Ασφαλείας και αναφερθήκατε και στην αναγκαία μεταρρύθμιση του ΟΗΕ διότι Γνωρίζουμε ότι η εκπροσώπηση της Ευρώπης δεν μπορεί να ρυθμιστεί με το να υπάρχουν ε, δύο μέλη μόνιμα ε, από την Ευρώπη στο Συμβούλιο Ασφαλείας που θα εγκαταλείψουν την ε, θέση τους αλλά η γερμανική έδρα θα μπορέσει να προσπαθήσει να γίνει μια ευρωπαϊκή έδρα κατά τρόπον ώστε να χρησιμοποιηθεί η Γερμανική Προεδρία κατά τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρηθεί σαν μια συνειδητοποίηση Ευρωπαϊκής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας πράγμα το οποίο θα συμβάλλει με τη, στην, στις διαβουλεύσεις με την Ευρώπη και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα μπορέσει να συμβάλλει στο να ενταθεί αυτή η συνειδητοποίηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω εν ονόματι των σοσιαλιστών να σας χαιρετήσω εδώ και χαιρόμαστε που διαθέσατε το χρόνο να κάνουμε μια εκτενή συζήτηση και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Συμφωνώ για τις ανάγκες μεταρρυθμίσεις στον ΟΗΕ. Ξέρουμε ότι αυτό δεν θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Θα είναι μια μακρά διαδικασία. Η συζήτηση δεν είναι καινούρια, αλλά τώρα πρέπει να δράσουμε και πρέπει να αναρωτηθώ και σε ένα θέμα πρέπει να επανέλθω στο, στη Λιβύη διότι ένα χρόνια, α, χρόνο μετά το ψήφισμα 1973 ε, α, αναρωτιόμαστε ε, εάν θα έπρεπε ε, να δύο μήνες, με συγχωρείτε, όχι δύο χρόνια. Μετά το ψήφισμα αυτό πρέπει να δούμε εάν έχουμε κινηθεί σωστά, αν έπρεπε να υπάρξουν οι σωστές προϋποθέσεις και αν αυτές δεν έχουν εξασφαλιστεί ε, και αν όλα τα θέματα δεν έπρεπε να έχουν διερευνηθεί πολύ περισσότερα. Δεν μπορώ να κρίνω σε αυτό το σημείο, αλλά σε μία δεύτερη τέτοια περίπτωση θα θα πρέπει να επιφυλαχθούμε γιατί αυτές ε, οι επαναστάσεις ε, δεν θα σταματήσουν και δεν μπορούμε να παραμείνουμε απλοί θεατές αλλά ε, δεν θα πρέπει να πάρουμε θέση στην λαθασμένη πλευρά του φράχτη. Παραδείγματος χάρη ο Καντάφη πρέπει να προσαχθεί σε ένα διεθνές δικαστήριο αλλά τότε θα λέγει ότι υπό αυτές τις προϋποθέσεις δεν φεύγω από τη Λιβύη και ε, σχετικά με την ε, εντολή του ΟΗΕ να προσάγει τον ε, Καντάφη στο διεθνές δικαστήριο επειδή είμαι εισηγητή σε μια επιτροπή για το θέμα αυτό, θα ήθελα να ακούσω ποια είναι η άποψή σας. Λάμστορφ, πρόεδρος και συντονιστής της ΑΛΔΕ και πρόεδρος της ομάδας εργασίας μας για τις σχέσεις με τα Ηνωμένα Έθνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είστε πολύ ευγενικός. Δεν είμαι όμως συντονιστής. Είμαι επικεφαλής της Υποεπιτροπής για τη σχέση με, την Ευρωπαϊκή, με τον ε, Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. πρέπει να σας πω ότι... Ε, υπάρχει η θέση ενός ε, κράτου τους ε, ε, που δεν είναι μόνιμο μέλος ε, του Συμβουλίου Ασφαλείας και εδώ πρέπει να συζητήσουμε με, τον, με τους Άγγλους και Γάλλους συναδέλφους αλλά και με τους Πορτογάλους επί του θέματος αυτού. Τώρα, η αντίληψη αυτή ότι η γερμανική θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας μπορεί να εκφραστεί σαν ευρωπαϊκή, τι σημαίνει συγκεκριμένα. Διότι από την πρώτη φορά που συζητήθηκε το θέμα το 2005 βλέπουμε ότι έχει γίνει μεγάλη πρόοδος όσον αφορά την πολυμορφία ε, ε, εις ε, το ψήφισμα 1970 ε, και 1973 στα ψηφίσματα αυτά βλέπουμε μία νέα διατύπωση είναι μία πρόοδος στον τομέα του διεθνούς δικαίου είναι ένας καλός ιονός για το μέλλον θεωρώ ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να συζητηθεί πέραν των πολιτικών ομάδων ε, και επίσης ε, πώς ασχολείται το Συμβούλιο Ασφαλείας με το θέμα της Συρίας, ε, πώς, ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Ο πρόεδρος Μεντβεντέφ έχει ήδη σχολιάσει το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να έχω περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Για να διευκρινίσω κάτι η κυρία Νέτση, συνάλφος Νέτση είναι συντονίστρια από την Άλντε. Μπουτικόφερα από του πράσινου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας χαιρετίζω κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο είναι ε, το πόσο θα επηρεάσει η γερμανική θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας το ψήφισμα 1973 και όπως είπε και ο κύριος ο Μπρόκ αυτό, αυτή η Προεδρία θα ακολουθήσει μία ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική διότι νομίζω ότι η έβαλε σε μεγαλύτερη απομόνωση της Γερμανίας και εντός της Ευρώπης διότι άκουσα στην Κίνα ότι η ομάδα BRIC έχει και ένα πέμπτο μέλος τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω πώς εσείς αντιλαμβάνεστε τη σημασία ε, της αρχής responsibility του protect, ευθύνη για προστασία διότι η απόφαση αυτή είναι πολύ σημαντική και πώς μελλοντικά ε, θα τη στηρίξετε ε, στη δραστηριότητά σας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Και μια δεύτερη ερώτηση. Πολύ σωστά είπατε κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών ότι εχθές αποφασίστηκαν σημαντικές κυρώσεις σχετικά με τη Συρία και τον πρόεδρο Ασάντ. Πριν δύο εβδομάδες δεν ήταν αυτό δυνατόν διότι ορισμένες χώρες είχαν αντιρρήσεις. Ε, ποιες ήταν αυτές οι χώρες και όντως εσείς πριν από δύο εβδομάδες ε, εμποδίσατε να ε, κατηγορηθεί ο Ασάντ. Τελευταίος ομιλητής του πρώτου γύρου, Λέζινγκ η συνάδελφος Λέζιν από την Ενωτική Αριστερά. Ευχαριστώ. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι αυτό το οποίο είπε ο κύριος Λάμσντοφ σαν διακομματικό δεν καλύπτει την δικιά μου θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Βέστερβέλ, πρώτη μου ερώτηση σχετικά με τη Λιβύη. Εσείς πιστεύετε ότι το ψήφισμα 1973 του ΟΗΕ είναι μία εντολή ε, για στρατιωτική αλλαγή του καθεστώτος όπως το έχουν εκλάβει ορισμένα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και αν όχι εσείς από δικιά σας άποψη ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι επιπτώσεις. Δεύτερο ερώτημα αναφέρεται εις ε, τις ε, έδρες στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μία θέση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Θεωρείτε ότι αυτή πρέπει να υπάρχει επιπλέον των δύο ισχυουσών ε, δρών και της μίας θέσεως που έχει ζητήσει η Γερμανία ή να υπάρχει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μία θέση που θα καλύπτει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και μία άλλη ερώτηση η οποία δεν αναφέρεται υποχρεωτικά στο θέμα αυτό αλλά το αναφέρατε στην αρχή και γι' αυτό επανέρχομαι. Κατά τη γνώμη σας ποιος είναι ο ρόλος του πολιτικού ιδρύματος αυτή τη στιγμή και εδώ αναρωτιέμαι ε, ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών ιδρυμάτων στην Αίγυπτο και άπαξ είσαστε εδώ θέλω να σας ε, ε, ρωτήσω το Ίδρυμα Νόρμαν τι ρόλο παίζει αυτή τη στιγμή στην Αίγυπτο. Κύριε Υπουργέ, ο λόγος ε, σε εσά. Θα ξεκινήσω κατά σειράν όπως με ρωτήσατε, συνάδελφε Μπροκ ε, η ευρωπαϊκή κοινή θέση στην, ε, ε, ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ είναι ο στόχος μας και θα είναι ο στόχος τον οποίο θα επιζητήσουμε μέσω της δραστηριότητάς μας για αυτή τη μεταρρύθμιση. Όπως σας είπα, η Λατινική Αμερική δεν εκπροσωπείται μόνιμα, η Αφρική δεν εκπροσωπείται μόνιμα, η Ασία είναι ε, ε, ε, υποεκπροσωπούμενοι δραματικά και σημαντικά και ε, εμείς ε, καλούμαστε να αναλάβουμε περισσότερες ευθύνες οπότε θεωρώ ότι η προσπάθεια ε, της Γερμανίας για μία θέση ήταν απλώς μία γέφυρα για να υπάρξει μία κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν θα εκπροσωπήσω δηλαδή τις γερμανικές θέσεις αλλά θέλουμε να συμβάλλουμε να ενισχύσουμε τον ΟΗΕ διότι εάν ο ΟΗΕ παραμείνει με τη μορφή που έχει τώρα θα χάσει τη σημασία του διότι εντωμεταξύ διαμορφώνονται νέα συστήματα τα οποία θα αναλαμβάνουν όλο και περισσότερες πρωτοβουλίες, θα λαμβάνουν όλο και περισσότερες αποφάσεις και θα πρέπει η κατάσταση του ΟΗΕ να αντικατοπτρίζει το σημερινό κόσμο. Βλέπουμε ε, όλο και περισσότερο παραδείγματο χάρη και εδώ δεν νομίζω ότι κομίζω γλάφκα στην Αθήνα ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να επιζητείτε. Ε, όσον αφορά τη θέση της Βραζιλίας η οποία όχι μόνο για ε, η δεν πρέπει να θεωρείται μόνο σαν μια οικονομικά επιτυχημένη χώρα αλλά θα πρέπει να αναβαθμιστεί και πολιτικά διότι ε, όταν μιλάμε για οικονομία μιλάμε για τα κράτη-μέλη μιλάμε για θέματα τα οποία μας απασχολούν εσωτερικά ενώ η πρόκληση για την Ευρώπη είναι να αντιμετωπίσει την δημογραφική εξέλιξη ανάπτυξη Δηλαδή οι περιοχές ιδιομογραφικά προηγμένες ε, σιγά σιγά θα ζητούν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή στα τεκτενόμενα όχι μόνο στα οικονομικά αλλά και στα πολιτικά και στα πολιτιστικά και σε όλα. Και δεν πρέπει να έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή εσωστρέφεια και να ασχολούμαστε τόσο λίγο με το τι γίνεται γύρω μας και εδώ για 50 χρόνια όπως γινόταν στο παρελθόν αλλά μέσα στα επόμενα 10 χρόνια θα συμβούν σημαντικές αλλογές οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν γίνονται αντιληπτές στην Ευρώπη και γι' αυτό θα πρέπει όλος ο κόσμος να έχει θέση στο Συμβούλιο Ασφαρίας. Και βέβαια δεν χρειάζεται εδώ σε τόσο εμπειρούς συναδέλφους να αναφερθώ τις δυσκολίες διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν μόνιμες θέσεις και δεν ε, σκέφτονται να εγκαταλείψουν τις ε, θέσεις τους αυτές. Δεν είναι τυχαίο ότι και οι πέντε παρεμβάσεις ήταν από Γερμανούς συναδέλφους ε, βλέπετε ποιος έχει συνέστηση της κατάστασης. Θα σας έλεγα όμως ότι το θέμα είναι πιο περίπλοκο και αναφέρεται σε περισσότερους. Δεν θα σας παρουσιάσω εδώ πολιτικούς στόχους, αλλά δεν ε, θα ε, αναφερθώ σε λεπτομέρειες τώρα. Είναι η τρίτη, τέταρτη συζήτηση που είχαμε τον πρόεδρο Ντάις, που είναι Ελβετός, και ε, βλέπετε ότι οι συζητήσεις δεν γίνονται μέσω του Γενικού Γραμματέα του Μπαν αλλά του Προέδρου ο οποίος δραστηριοποιείται σε αυτή τη μεταρρύθμιση των δομών. Επαναλαμβάνω λοιπόν εδώ μέσα ότι ο στόχος μας ε, για τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ δεν είναι να υπάρχει μεγαλύτερο ε, εθνικό βάρος αλλά να υπάρξει μία μεταρρύθμιση των δομών και οι Γερμανοί θεωρούμε ότι πρέπει να προετοιμάσουμε μία μοναδική ευρωπαϊκή εκπροσώπηση. Ε, κύριε συνάδελφε, ε, κατακρίνατε την ε, θέση της Γερμανίας στην ψηφοφορία, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν τη συμμερίζομαι την θέση αυτή, διότι πιστεύω ότι ήταν μία πολύ δύσκολη απόφαση και πιστεύω ότι τελικά ήταν η σωστή απόφαση αυτή στην οποία καταλήξαμε. Διότι από την αρχή θέσαμε το βάρος σε μία πολιτική αλλαγή και πιστεύουμε ότι η στρατιωτική παρέμβαση πρέπει πάντοτε να μένουν η ίστατη λύση και για μένα είναι ένα αποτύπωμα της εξωτερικής μου πολιτικής να ακολουθήσω ε, ε, την γερμανική άποψη. Δεν επαρκεί σαν Γερμανός υπουργό των Εξωτερικών να λέω στο κοινοβούλιο μας ότι συμμετέχουμε σε ε, στρατιωτικές επεμβάσεις γιατί το κάνουν άλλοι ακόμη και αν είναι οι καλύτεροι μας φίλοι πρέπει εμείς να είμαστε πεπισμένοι για, την, για τις ενέργειές μας. Ε, όσον αφορά τα, ε, ε, τις υπόλοιπες υποθέσεις οι οποίες αναφέρθησαν δεν θα τις σχολιάσω αλλά ξέρετε ο κύριος, ξέρετε ο κύριος Στάιν Μάιερ πώς συμπεριφέρθηκε ο, ο οποίος αξιολόγησε και επένισε την αποχή μας δεν θέλω λοιπόν να δώσω την εντύπωση ότι υπάρχουν διαφοροποιημένες θέσεις εσωτερικά στη Γερμανία. Ε, εάν ε, ε, είχα δώσει αυτή την εντύπωση τη διασκέδασα τώρα. Επίσης, στόχος μας είναι κύριοι συνάδελφοι ο, ο Καντάφη και οι συνέτεροι του να καταλήξουν στο δικαστήριο αυτό είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας και είναι ο πυρήνας της πολιτικής διαδικασίας που ακολούθησε η Γερμανία. Και το επαναλαμβάνω προς τους άλλους συναδέλφους άλλων χωρών. Σέβομαι όποιος με, ε, με διαφορετικά κίνητρα κατέληξε σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Εγώ όμως είμαι πεπισμένος ότι η Γερμανία το αργότερο τώρα θα είχε καταλήξει σε μια διαφορετική συζήτηση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι βλέπουμε τι σημασία έχει ε, η στρατιωτική επέμβαση και η ε, ομάδα επαφών για τη Λιβύη όπως συμμετέχουμε όπου πάντοτε τονίζεται η ανάγκη μιας πολιτικής διαργασίας και αν διάβασα σωστά τα ψηφίσματά σας συμμερίζεστε την άποψή μου. Οπότε ε, ε, δεν πιστεύω επιπλέον ότι πρόκειται για μία έξυπνη πολιτική να θεωρήσει κανείς ότι μία περίπτωση αποτελεί προηγούμενο για άλλες περιπτώσεις. Δηλαδή όταν μου λέτε τι θα κάνατε σε συγκρίσιμες περιστάσεις. Θεωρώ ότι αυτό είναι λάθος αντιμετώπισης. Εγώ δεν θα συμμετάσχω σε τέτοιες συζητήσεις διότι αυτή η γενίκευση της ε, επανάστασης στη Βόρειο Αφρική είναι μια γενικευση με το σύνθημα ότι η Λιβύη, η Συρία, η Εμέν, το Μπαχρέιν και ίσως το Ιράν. Αλλά αγαπητοί συνάδελφοι, η κατάσταση διαφέρει πάρα πολύ από τη μια περίπτωση στην άλλη. Συγκρίνουμε ε, δύο μοναρχίες οι οποίες εξελίσσονται διαφορετικά, η Ορδανία και το Μαρόκο. Ακόμη και αν αναφερθείτε εις ε, την ε, θρησκευτική αρχή του Μοχάμε του Έκτου, ο οποίος από την αρχή επέβαλε μία πολιτική μεταρρύθμιση με την οποία δεν συμφωνούσαμε, η οποία όμως ξεκίνησε. Διότι μίλησα με την αυτού υψηλότητα προημερών και μου είπε ότι επιθυμεί μεταρρυθμίσεις. Αυτό, είναι το... Αυτό σημαίνει σωστή πολιτική και γι' αυτό δεν μπορώ μετά από μία στρατιωτική επέμβαση σε μία χώρα να προεξοφλήσω ότι το ίδιο πρέπει να γίνει σε μία άλλη χώρα και δεν νομίζω ότι το ίδιο συζητούν οι σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη. Αυτό θα με ανησυχούσε. Ε, κάποιο σχόλιο που δεν ακούστηκε. Ναι, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το δύσκολο. Και πάλι δεν θέλω ε, να σας αλλάξω γνώμη, αλλά εγώ δεν ε, μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας. Μπορούμε να έχουμε καλά αποτελέσματα και με διαφορετικές μεθόδους. Όσον αφορά τον ΟΗΕ, ε, θα ζητούσα να, κοιτάξουμε με τους συναδέλφους να ασχοληθεί ε, ε, ο και το Συμβούλιο Ασφαλείας με τη Συρία αλλά υπάρχουν παντού ορισμένοι εταίροι οι οποίοι είναι πολύ πιο επιφυλακτικοί δεν χρειάζεται να σας το εξηγήσω τώρα οπότε πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν στη συνέχεια τα θέματα αυτά αλλά η ουσία είναι σωστή και βεβαίως όσον αφορά την responsibility του protect θεωρούμε ότι είναι βασική πρόοδος αλλά responsibility to protect δεν σημαίνει να κατεβάσουμε τον πύχη για την παρεμβατικότητα διότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Responsibility to protect θα πρέπει να προσανατολίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια και δεν πρέπει να μειώσει τον πύχη για τις παρεμβάσεις διότι από τις καλές προθέσεις μπορεί να έχουμε πολύ κακές και δύσκολες επιπτώσεις. Έχω απαντήσει στα περισσότερα τα οποία είπατε συνάδελφοι. Δεν αντιλαμβάνομαι καταρχήν. Βεβαίως με ενδιαφέρουν τα νέα σας από την Κίνα και τον αναφέρεστε εδώ στην Κίνα διότι και εκεί η responsibility του protect είναι μία αξιέπαινη διαδικασία. Εσείς πρέπει να ντραπείτε για τους εταίρους σας στη συμμαχία, όχι εγώ λέει ο κύριος Μπιτικόφερ. Δεν ε, καταλαβαίνω τι εννοείται με αυτό γιατί μιλήσατε για απομόνωση στην Ευρώπη και πρέπει να σας πω ότι τα, ε, περισσότερα κράτη της Ευρώπης δεν συμμετείχαν, σε δεν συμμετείχαν στρατιωτικά. Είναι βέβαια δικιά σας ε, απόφαση να στηρίζετε την στρατιωτική ενέργεια. Εγώ παρουσίασα τις δικές μου απόψεις και ε, εάν η, αυτή είναι η πράσινη πολιτική για την Ευρώπη θα το μεταφέρω στη χώρα μου. Αλλά ε, όσον αφορά τη Συρία Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αποφασίσει να προχωρήσουμε σε δύο, σε ε, στάσεις. Δηλαδή πρώτα θα υπάρξει ένας κατάλογος απαιτήσεων για τη Συρία και αν δεν καλυφθούν τότε θα ζητήσουμε κυρώσεις κατά του Προέδρου Ασάντ και ξέρετε ότι ε, αυτά τα μέτρα ελήφθησαν. Εχθές ελήφθη μια σημαντική απόφαση. Κυρία Λέζινγκ, ε, θα αναφερθώ σε ένα θέμα, για τα υπόλοιπα τα έχω απαντήσει από αυτά τα οποία είπατε. Με συγχωρείτε ε, και θα, ε, δεν μπορώ εδώ να αναφερθώ σε, μία, σε ένα ίδρυμα, το Ίδρυμα Φρίντριχ Νόημαν, διότι έχω συζητήσει με τους εκπροσώπους όλων των γερμανικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται πολύ καλά στην κοινωνία των πολιτών και ενθαρρύνω όλα τα ιδρύματα να χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες να παρέμβουν στις χώρες δημοκρατικών εξελίξεων και να επηρεάσουν την κατάσταση. Πιστεύω ότι είναι καλός χώρος για τα ιδρύματα αυτός, ιδίως όταν κατευθύνονται πολιτικά από τη χώρα προελεύσεώς τους δεύτερος γύρος. Πολλοί έχουν ζητήσει το λόγο, γι' αυτό ένα λεπτό μόνο δυστυχώς ε, χρόνος ομιλίας για τον καθένα. Ο συνάδελφος Αλαφράνκα πρώτος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Υπουργέ γιατί σήμερα είστε εδώ. Δεν είμαι Γερμανός, πάντως ε, είδα ότι η ψήφος της Γερμανίας ε, ήταν αποχής. Έχω όμως μέσα αμφιβολίες ότι είναι θετικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτά τα λίγα μέλη μας στην, ε, στο Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να ψηφίζουν ομόφωνα. Αυτό λοιπόν ελπίζω ότι θα προσπαθήστε πάντως για κάτι καλύτερο. Η Γαλλία αρκετές φορές θέλησε να έχουμε ένα ειδικό απεσταλμένο για την ε, για τη Μεσανατολή. Αλλά κύριε Άστον δεν θέλησε μέχρι να τελειώσει ο ρόλος του κύριου και η εντολή του κύριου Μπλερ. τι φρονείτε εσείς η χώρα σας και για τη Λατινική Αμερική ότι δεν έχει μόνιμη θέση στο Σύμβολο Ασφαλείας. Τι γίνεται με αυτό. Η Γερμανία όμως υποσχέθηκε ε, για την, ε, να αποδεχτεί αυτό που έγινε τώρα και με την κυρία Βάγνερ και πρώτη πρόεδρο αυτού του Ιδρύματος με έδρα το Αμβούργο. Υπάρχουν προβλήματα σχετικά με το νομικό καθεστώς του Ιδρύματος σύμφωνα με το γερμανικό δίκαιο. Εσείς ε, λέτε ότι θα υποστηρίξετε αυτό το Ίδρυμα και πώς έχει κατάσταση, ποια προβλήματα υπάρχουν και πώς θα δοθεί ένας δυναμικός χαρακτήρας για να μπορέσει να παίξει ενεργό ρόλο το Ίδρυμα αυτό ανάμεσα σε αυτές τις περιοχές. Вигени από τους σοσιαλιστές. Κύριε Βεστερβέλα, χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που μπορούμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας για ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το ρόλο της Γερμανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Θα ήθελα δύο σχόλια να κάνω πριν ε, θέσω και την ερώτησή μου. Καταρχάς, πιστεύω ότι Κάνετε λάθος όταν λέτε ότι η Γερμανία θα έπρεπε να αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο γιατί είναι και μεγαλύτερος χρηματοδότησης. Κοιτάξτε, Υπάρχουν πολλές χώρες οι οποίες ε, μπορεί να ε, έδιναν ακόμη περισσότερα χρήματα. Πρόκειται για ένα ρόλο τον οποίο θα μπορούσαν ε, να έχουν και άλλες χώρες, θα μπορούσαν να δώσουν πολύ περισσότερα. Εμείς πιστεύουμε ότι ε, η Γερμανία δεν συμμετέχει επαρκώς ε, στις ε, ισχυρές δεσμεύσεις που έχουν αναλυφθεί και αν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε μία έδρα ε, μήπως θα αργούσαμε πολύ περισσότερο γιατί δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε επί συγκεκριμένων ζητημάτων πολύ γρήγορα. Ποια είναι η άποψή σας για, την για τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο πλαίσιο του ΟΗΕ. Επίσης υπάρχει ένα ζήτημα για το οποίο εσείς προσωπικά θα θέλατε η Γερμανία να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο, όπως για παράδειγμα το θέμα της Κύπρου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε. Δεν είμαι Γερμανός ή Γερμανόφωνος, αλλά για να μην νομίζετε ότι βρίσκεστε στο Γερμανικό Κοινοβούλιο, θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου που είναι Σλοβένικα. Δυστυχώς υπάρχει ένα κάποιο πρόβλημα στη Γερμηνία. Μισό λεπτό παρακαλούμε. είναι, είναι ε, Παρακαλώ. Κύριε Βάγγελ, μήπως θα μπορούσατε να χρησιμοποιείτε και πάλι γερμανικά για να σας καταλάβουμε έτσι. Ich kriege eine Ermäßigung, wenn es um Zeit geht dann, τότε με συγχωρείτε αλλά δώστε μου περισσότερο χρόνο διότι στις δύο τελευταίες ομιλίες του Αμερικανού Προέδρου ε, αντιληφθήκαμε ε, την, ε, το βάθος και τις περιπλοκές του προβλήματος της Μέσης Ανατολής όπου εξετάστηκαν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που ανοίγουν και επιπρόσθετα θέματα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω το εξής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία διότι αυτή τη στιγμή δεν διαδραματίζει κανένα ρόλο. Ε, όπως ε, το, όπως άλλωστε διαπίστωσαν και άλλοι παλαιοί ειδικοί διαπραγματευτές. Εσείς λοιπόν πώς ε, εκλαμβάνετε την ε, ε, συμμετοχή σας ή το Συμβούλιο Ασφαλείας επί του θέματος αυτού και έτσι κάλυψα όλο μου το χρόνο. Πολύ καλά λέει ο Πρόεδρος. Και πάλι γερμανικά. Σούλτς. Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών Βέστερβέλε, αυτή τη στιγμή διεθνώς και εθνικά δεν σας επενούν πολύ και εγώ θα επανέλθω στην τριμερή συζήτηση στο Καλίνιγκραν ε, που φέρει το όνομα ενός ε, σταλινιστή που ενεπλάκει στη σφαγή του Κατίν. Ε, βλέπω ότι υπήρξε αυτή η συζήτηση τριμερής και δημιούργησε μία ε, ε, ελπίδα για το θέμα της Τρανσνιστρίας ε, επί του οποίου όμως δεν έχω ακούσει εξελίξεις εδώ και πολύ καιρό και θα ήθελα να ξέρω που βρίσκεται. Κόβατσεφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ που ήρθατε εδώ. Η Ευρώπη δίνει την περισσότερη βοήθεια και ανθρωπιστική βοήθεια παντού ανά τον κόσμο όσο θέλω και να σεβαστώ το πολιτικό βάρος της Ευρώπης. Όμως πιστεύω ότι σε αυτό είμαστε ακόμη πολύ μικροί και δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κοινή πολιτική γραμμή στην Ευρώπη. Όσον αφορά την και την αποδοχή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από τους διεθνείς οργανισμούς είναι για μας ένα σημαντικό θέμα και από αυτού θα ήθελα να ξέρω πώς συνεργάζεστε με την Ευρωπαϊκή Εξωτερική Υπηρεσία και με την κυρία Άστον για να πετύχετε αυτό το στόχο και για να μπορέσει η Ευρώπη να επεμβαίνει όλο σε περισσότερα θέματα ε, διότι θα θέλαμε στο μέλλον να αποφεύγουμε τις εκπλήξεις εθνικών ε, αντιλήψεων και στο τέλος ε, πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ότι ε, ε, στη Γερμανία συζητείται ακόμη ε, το θέμα του Ευρωπαϊκού στρατού. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν τι κάνει η Γερμανία επί του θέματος αυτού εφόσον ούτως ή άλλως η Γερμανία είναι ο κινητήρας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Από πλευρά σοσιαλιστών Αντιπρόεδρος Πασκού. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ένα από τα αποτελέσματα της τρέχουσας κρίσης είναι το γεγονός ότι μας κάνει να ενδοσκοπούμε περισσότερο, να είμαστε λίγο πιο εσωστρεφείς και να κρίνουμε όχι ως ε, τέτοια τα διεθνή ζητήματα, αλλά βάσει του αντικτύπου που έχουν ε, στην ε, κοινή γνώμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το προφανές και είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη συνοχή και την συντονισμένη ανταπόκριση που θα θέλαμε μερικές φορές να έχει. Την επόμενη χρονιά έχουμε εκλογέ σε πολλέ σημαντικέ χώρε ε, και στην Ευρώπη αλλά και εκτό Ευρώπη. Ε, θα έχουν είτε βουλευτικέ είτε προεδρικέ εκλογέ και υπό τι συνθήκε αυτέ αναρωτιέμαι κατά πόσο είστε πιο ε, αισιόδοξο ή απεσιόδοξο σε σχέση με τα αποτελέσματα των εκλογών αυτών στα διεθνή ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μπράντνερ από πλευράς Πρασίνων. Κύριε Υπουργέ Εξωτερικών Βέστερ Βέλε, σχετικά με τη Λιβύα, μιλήσατε για μια διαδικασία, αλλά ποια είναι η συγκεκριμένη πρότασή σας, μπορείτε παρακαλώ να μας την διευκρινίσετε και όσον αφορά την Βόρειο Αφρική και την Αίγυπτο, συναντηθήκατε με το Διεθνές Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο ε, ε, είχε ανανεώσει τη συμμετοχή του, αλλά πάλι πρόκειτο για ανδρίκελα των κυβερνήσεων και όχι για ανεξάρτητα άτομα οπότε γιατί επικυρώνετε την εκλογή του με την συμμετοχή σας ε, γιατί λοιπόν χρηματοδοτείτε και ενθαρρύνετε την ε, χορήγηση θεωρήσεων για αυτές τις χώρες είναι και ε, σχετικά με το ε, ψήφισμα 1325 του ΟΗΕ. Τι γίνεται. Και τέλος ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ. Παρόλες ε, τις σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή παραμένει το θέμα αυτό οξύ και σχετικά με τη, τα τελευταία σχόλια του Αμερικανού Προέδρου στους τελευταίους λόγους του σύμφωνου με τις απόψεις τους για την επαναφορά των συνόρων του 1967 και πώς αυτό θα μας επηρεάσει ε, στην Ευρώπη και ε, με την Προεδρία της Γερμανίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ε, πιστεύετε ότι η πολιτική ένωση των Παλαιστινίων είναι εφικτή και είναι μία συμμετοχή η οποία θα διευκολύνει ή θα, διευ... Ε, ή θα καταστήσει πιο δύσκολη την επίλυση του προβλήματος της Παλαιστίνης. Επίσης, ε, όσον αφορά ε, τις εγκαταστάσεις στη Δυτική Όχθη, ε, τι γίνεται, δεν πρέπει κανείς να πιέσουμε το Ισραήλ αν υπάρχουν αποφάσεις οι οποίες λαμβάνονται ενάντια προς, προς τα διεθνή ψηφίσματα. Ευχαριστώ για την απάντηση τώρα ο κύριος Βεστερβέλε σχετικά με το Ίδρυμα της ε, ε, Λατινικής Αμερικής. Πιστεύουμε ότι με το Ίδρυμα αυτό ε, θα έχουμε ένα σημαντικό οργανισμό στο Αμβούργο. Συζήτησα το θέμα με τη νέα πρόεδρο και την Γενική Γραμματέα διότι έχουμε ακόμη διάφορες δυσκολίες. Υποθέτω ότι το γνωρίζετε και γι' αυτό κάνατε την ερώτηση. Το προτεραιότητας είναι πότε θα ξεκινήσει δουλειά αυτός ο οργανισμός. Νομίζω ότι σας είπα τι γίνεται, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη νομική μορφή για να μπορέσει να ξεκινήσει αυτή η οργάνωση Υπάρχει και ένα ποσό το οποίο έχει διατεθεί ε, σχεδόν 300.000 ευρώ το οποίο είναι ε, ε, καλό για ένα ξεκίνημα και σε σχέση με τις σχέσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής θα έχει μεγάλο σημαντικό θα έχει μεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον για τις σχέσεις με τη Βραζιλία που ήδη προανέφερα αλλά παραδείγματο παραδείγματος χάρη ε, και για τις επισκέψεις ε, ε, της την επίσκεψη του Προέδρου εις ε, τη Λατινική Αμερική προμίας εβδομάδος διότι λέμε ότι οι Ισπανοί, οι Πορτογάλοι έχουν δημιουργήσει μια πολύ ισχυρή γέφυρα προς τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκό ενδιαφέρον όχι μόνο για πολιτιστικούς λόγους αλλά και για στρατηγικές σκοπιμότητες πέραν των οικονομικών ε, αναφερθήκατε επίσης για τον ΟΗΕ, το στηρίξαμε, ήταν η πολιτική μας από την αρχή. Θέλαμε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια αυτή και θα την συνεχίσουμε. Ε, κύριε συνάδελφε, αναφερθήκατε ή κάνατε το ερώτημα για την ε, απέτηση της Γερμανίας για μία θέση μόνιμη στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Αλλά εμείς με αυτόν τον τρόπο προσπαθούμε να αναλάβουμε πολλές πολιτικές ευθύνες ε, και πέραν των καταβολών των συμμετοχών που δεν είναι πουσιώδης. Ε, πιστεύουμε ότι η διεθνής ευθύνη ε, δεν πρέπει να αξιολογηθεί μόνο από στρατιωτική σκοπιά, αλλά πρόκειται για διασύνδεση, για την εφαρμογή ειρηνικής πολιτικής, και η ε, Γερμανία ενδιαφέρεται για την αναπτυξιακή συνεργασία ε, με τις υποανάπτυξη χώρες και ε, πιστεύουμε ότι η Γερμανία είναι μια χώρα που μπορεί να συμβάλλει θετικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας σε πολλαπλά θέματα. Όσον αφορά τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην ειρηνευτική διαδικασία της Μέσης Ανατολής, προφανώς πρόκειται για ένα από τα πιο δύσκολα θέματα και έχει σχέση με αυτό το οποίο αναφέρθηκε και στο τέλος σχετικά με ε, τα σύνορα που ε, προαναφέρατε. Ο ρόλος της Ευρώπης στη διαδικασία την ειρηνευτική της Μέσης Ανατολής από όταν αναβιώσαμε ε, το κουαρτέτο με την διακήρυξη της Μόσχας πρέπει να ενισχυθεί. Ε, διότι η τετραμερής αυτή προσπάθεια ε, έχει αποδώσει και το διαπιστώνουμε. Ε, υπάρχει μία άμεση συζήτηση μεταξύ των εμπλεκομένων για ειρήνευση και σε αυτό συνέβαλε ο πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος δεν ζήτησε να επανέλθουμε στα σύνορα του 1967, αλλά στα σύνορα αυτά με συμπεφωνημένες ανταλλαγές γεών with agreed land swaps και ε, αυτό συμμετέχει στην απόφαση και όποιος το ξεχνά δεν ε, ε, αξιολογεί σωστά την κατάσταση για τους Ευρωπαίους αυτό δεν είναι μία ε, ε, θεαματική αλλαγή τοποθετήσεως διότι εάν λάβετε υπόψη την πρωτοβουλία του Φεβρουαρίου στο Συμβούλιο ε, Ασφαλείας για την πολιτική επικίσεως στη Δυτική Όχθη είχα συζητήσει το θέμα αυτό και με τους Βρετανούς και ψηφίσαμε από κοινού κοινού, η Ευρώπη ψήφισε όλοι από κοινού, αλλά αντιμετωπίσαμε το βέτο των Ηνωμένων Πολιτειών η επική ε, ε, δεν είναι κάτι νέο για μας τους Ευρωπαίους και το έχω συζητήσει αυτό και στο Ισραήλ. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν είναι σωστό να υπάρξουν μεμονωμένες κινήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να τις εγκαταστήψουμε. Ο κύριος Σούλτς μίλησε για το Καλίνιγκρακ. Ναι, το συζητάμε, είναι δύσκολο θέμα, αλλά το θίγουμε, μιλάμε και για την Τρανσνιστρία. Η συζήτηση 5 επί 2 μπορεί να ξαναξεκινήσει τώρα και με τον ε, Υπουργό Εξωτερικών Λεάνκα ε, της ε, Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Συζητήσαμε προημερών στα πλαίσια του τριγώνου της Βαϊμάρης και είμαι ο πρώτος Υπουργός Εξωτερικών ο οποίος επισκέφτει τη Μολδαβία και θεωρούμε ότι δεν είναι μόνο θέμα της πρωτοβουλίας του Μέζενμπεργκ αλλά είναι ευρωπαϊκό μέλημα. Πρέπει να ανησυχούμε. Ε, δεν πρέπει να μιλάμε για frozen ε, ε, conflicts αλλά για frozen solutions και πρέπει να τις προωθήσουμε τις λύσεις αυτές. Άκουσα τι θέματα έχει θίξει η συνάδελφος Άστον και πρέπει να σας πω ότι όλοι οι οποίοι μιλούν για αυτή την υπηρεσία πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή πόσο ε, δημιουργήθηκε και καταρτίστηκε η εξωτερική αυτή υπηρεσία. Δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολα και πρέπει να μιλάμε για τις επιτυχίες. Αναφέρθηκα στον ΟΗΕ αλλά υπάρχουν και άλλα διότι ε, ε, πέρυσι η πρωτοβουλία του William Hague για τη Σερβία, το Κωσυφοπαίδιο και τη σχετική ψηφοφορία στον ΟΗΕ είναι μια πρωτοβουλία χαλαρώσεως την οποία αναλάβαμε πέρυσι το καλοκαίρι με τον William Hague και η προσπάθεια αυτή έχει συνδυαστεί με τις έξυπνες κινήσεις ε, και δηλώσεις της ε, Ladies Ashton και άρα θεωρώ ότι είναι θετική η συμμετοχή της. Και όταν κάνουμε ε, επισκέψεις σε χώρες κύριε Πάσκου ε, μπορεί να μιλάμε με πολλούς οργανωμένους εκπροσώπους και με προσωπικότητες οι οποίες δεν είναι οργανωμένες και πρέπει να σας πω ότι η επιρροή της Γερμανίας και η πολιτική της Γερμανίας εις την Αίγυπτο έγιναν αποδεκτές θετικά όπως και στην Ισία χωρίς να συνεπάγεται αυτό ότι δεν στηρίζουμε την προσπάθεια αυτή την οποία προσπαθούμε να ενισχύσουμε και οικονομικά. Και τέλος θα μιλήσω αγγλικά. Καταλαβαίνω την ανησυχία σας και νομίζω ότι έχετε απόλυτα δίκιο όταν λέτε ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή προσανατολίζεται πάρα πολύ σε ε, εσωτερικά ζητήματα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις από κοινού και με άλλα, άλλες περιοχές του κόσμου. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που προσπαθώ να ε, πω κι εγώ. Δεν θα ήθελα να υπάρχει καμία αμφιβολία αν υπάρχει κάποια αμφιβολία και έτσι το διαισθάνομαι αυτό πίσω από αυτά που είπατε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν αμφιβολίες για την γερματική δέσμευση σε σχέση με την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μας ε, για μας αυτό είναι και επιθυμία, αλλά είναι και το πεπρωμένο μας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και αν έχω, την, ε, το, αν έχω το προνόμιο να το πω αυτό και σε χώροι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορώ να το πω και σε εσά. Το μέλλον της Γερμανίας είναι στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν διαπραγματεύσεις αλλά για τη γερμανική εξωτερική πολιτική είναι σαφέστατο ότι η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ευρωπαϊκό συμφέρον, είναι και εθνικό μας συμφέρον αν θέλουμε να έχουμε μια καλύτερη ζωή για τους λαούς μας στο μέλλον και κυρίως για τους νέους, για τις νεότερες γενναίες. Και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να αποδεχθούμε καμία συζήτηση για επανεθνικοποίηση, η απάντησή μας ε, στα κράτη-μέλη μας ε, δεν μπορεί να είναι μια απάντηση επανεθνικοποίησης, ε, για παράδειγμα παρεμπόδιση ε, των ε, δικαιωμάτων ε, ελευθερίας της κυκλοφορίας, για παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω να έπεισα τους Ευρωπαίους συναδέλφους που θα συμμετέχουν στις συζητήσεις μαζί μας δεν υπάρχει καμία ανάγκη. Ενδεχομένω υπάρχουν κάποιες φήμες σε κάποιε πρωτεύουσες αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει δεν, δεν υπάρχει ε, κανένας λόγος να πιστεύετε ότι δεν θα είμαστε αρκετά συνεργάσιμοι ως Γερμανοί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ε, θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκαταλείψει το κτίριο σε 11 και 4 ο κύριος Υπουργό. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω και από μέρους μου και από τον συνάδελφο Ντονζάν. Μήπως θέλει κάτι να προσθέσει. Όχι. Σας ευχαριστώ. Η παρουσίασή σας ήταν πολύ πολύ καλή. Αγαπητοί συνάδελφοι, επανερχόμαστε στις εργασίες μας για την υποεπιτροπή μας. Παρακαλώ στις θέσεις σας όλοι, σας ευχαριστώ. Και στη μέση μας διάταξη έχουμε ένα τελευταίο μέρος που έχει να κάνει με την παρέμβαση του κ. Ντεκερκόφ, συντονιστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Θα θέλαμε να σας ευχαριστούμε για την υπομονή που επιδείξατε, γιατί καθυστερήσαμε κάπως. Ε, έρχεστε αρκετά συχνά εδώ στην Επιτροπή μας, σας ευχαριστούμε και σήμερα αυτά που θα πείτε έχουν να κάνουν με τις πρόσφατες εξελίξεις ε, για την Αλκάιντα και τέλος του Μπιν Λάντεν. Θα θέλαμε να ακούσουμε τη δική σας την εκτίμηση, τι λέτε σχετικά. Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, επειδή ήδη σημαίνει μια καθυστέρηση, γι' αυτό σας παρακαλώ στις θέσεις σας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, αυτό με τον Μπεν Λάντεν, τι γίνεται, ποιε είναι συνέπειες, σύμφωνα με αυτά μπορεί να κρίνετε εσείς επιχειρησιακά για την Αλκάιντα και επιχειρησιακά επίσης και για άλλα κινήματα γύρω από αυτήν όπως το Ισλαμικό Μαγκρέμπ που ε, έχουν πάντα διάφορους ομήρους ε, και διάφορα αυτά τα πρόσφατα στο Μαρακές ε, και νομίζω ότι η πείρα σας ιδιαίτερα θα μας ωφελήσει εδώ και ακόμα για τη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε σίγουρα δεν μπορείτε να μας αποκαλύψετε πράγματα για ευαίσθητου τομεί, αλλά μετά από αυτό που έκανε οι Αμερικανοί στο Πακιστάν, την επέμβασή του, έχουμε την δυνατότητα με του Αμερικανού να δούμε με ποια μέθοδο μπορούμε να δούμε κάτι σχετικά με αυτή την επιχείρηση, μετά από διάφορα που ακούσαμε εδώ και φήμε εδώ και εκεί, για διάφορε παρεμβάσει ε, όπω σχεδιάστηκαν, την παρέμβαση που σχεδιάστηκε σε κράτη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τι γίνεται ακριβώ, μετά από αυτό που συνέβη με τον Μπελάντεν και επίσης από πολιτικής πλευράς το ότι ο Μπελάντεν ε, ήταν ε, ε, κατά τις συνθήκε που γνωρίζουμε στο Πακιστάν. Τι γίνεται αυτό, επηρεάζει τα πράγματα στο διάλογό μας με το Πακιστάν για θέματα ασφάλειας και αντιτρομοκρατίας. Είναι σημαντικά αυτά τα θέματα, θα θέλαμε να τα εξετάσουμε μαζί σας και ακόμα έτσι οργανωτικά ακριβώ επειδή εσείς ε, έχετε σχέση με αυτά, τι γίνεται μετά από Λισαβόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς λειτουργούν ε, οι εξωτερικές υπηρεσίες της Επιτροπής και εσείς ε, στα πλαίσια αυτά τι θέση κατέχετε. Καλό θα ήταν να τα ακούσουμε όλα αυτά 1,5 χρόνο μετά από τη θέση ισχύ της ε, συνθήκης και ενδεχόμενα και συνάδελφοι θα έχουν περαιτέρω ερωτήσει να σας απευθύνουν. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ κάθε φορά που, πρέπει, που έρχομαι στην ε, συγκεκριμένη επιτροπή ε, και κάθε φορά μου δημιουργείται μεγάλος προβληματισμός μετά από τις συζητήσεις μας. Τρία σημεία θα ήθελα να θέσω και όπως είπατε και εσείς, ε, τον, τον αντίκτυπο του θανάτου του Οσάμα Μπιν Λάντεν και θα ήθελα επίσης και τις συνέπειες, να συζητήσουμε τις συνέπειες της Αραβικής Άνοιξης στην τρομοκρατική στην αντιτρομοκρατική δράση. Υπήρξαν μέχρι την, από την τελευταία μα ε, συζήτηση πολλέ ενδιαφέρουσε εξελίξει και υπάρχει, και υπάρχει το θέμα που θέσατε εσείς, ε, το θεσμικό περιβάλλον και πώ μπορούμε να κινητοποιήσουμε κάθε καλή θέληση, κάθε πόρο, κάθε μέσο για να έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της ε, απειλής κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο ζήτημα που θα ήθελα να θέσω συζητήθηκε και από τους 27 Υπουργούς Εσωτερικών την περασμένη εβδομάδα έφτασαν ε, στο συμπέρασμα και εγώ συμμετείχα σε αυτές τις συζητήσεις. Καταρχάς, ο θάνατο του Οσάμα Πινλάντε ήταν ένα τεράστιο θέμα στι ΗΠΑ. Πολιτείε. μια μεγάλη επιτυχία για όλου, για όλους όσους ε, ε, είχαν επενδύσει προσπάθειε προσπάθειες ε, στην αντιτρομοκρατική δράση. Από, από πολιτικού συμβολισμού είχε ήδη πεθάνει κατά κάποιο τρόπο ο Σάμα μέσω όσων έγιναν κατά την Αραβική Άνοιξη, γιατί όλοι αυτοί ε, ό, όλος αυτός λόγος ε, που χρησιμοποιούσε ο Σάμα Μπιν Λάντεν φαινόταν ότι δεν είχε πλέον κανένα αντίκτυπο. Ήταν λοιπόν ένα θετικό, ήταν θετικός ο αντίκτυπος ε, στον ε, αραβικό κόσμο γιατί ε, οι περισσότερες τρομοκρατικές οργανώσεις μουσουλμανικές που εμπνέονται από την Αλκάιντα ε, έχουν πλέον αποδυναμωθεί και πολύ συχνά μάλιστα υπήρχαν σχέσεις με το Πακιστάν. Είναι πολύ νωρίς ε, για να πει κανείς και απαντώ εμέσως ε, στο ερώτημά σας ε, σε σχέση με το θησαυρό αυτό που, είχαμε, που βρήκαμε στο Αμπούνταμπάντ για να δούμε ακριβώς πολλά επιχειρησιακά στοιχεία του Σάμα Μπιν και της Αλκάιντα. Ε, ούτως ή άλλω θα γίνει και διάλογος με τους Αμερικανούς για το θέμα αυτό κατά τις επομενε δυο δύο-τρει εβδομάδες και είμαι σίγουρος ε, ότι σε επιχειρησιακό επίπεδο θα αναφερθούμε κυρίως στο κατά πόσο συμμετείχε άμεσα στη, στο σχεδιασμό των ε, επιθέσεων. Ξέρετε ότι υπήρξαν συλλήψει στον Ντίσελντορφ προσφάτω και αυτό είναι κάτι που παρακολουθεί το από τον ίδιο τον Οσάμα Μπιν Λάντεν. Μιλήσατε για τις απειλές κατά τρένων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, θα ήθελα να επαναλάβω μάλιστα αυτό που λέω κάθε χρονιά, αλλά μέχρι τώρα δεν είχα εισακουστεί ότι είναι ενδεχομένως ε, ο τομέας των μεταφορών για τον οποίο θα έπρεπε να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο, δηλαδή τα τρένα ταχείας ε, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και είναι πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν οι απειλές σε σχέση με τι απειλέ στις θαλάσσιε μεταφορέ και σε αεροπορικέ μεταφορέ. Πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε δηλαδή ε, την ε, ασφάλεια του τομέα αυτού μεταφορών ε, και στι μεγάλε πόλει. Υπάρχει λοιπόν ιδιαίτερη, υπάρχουν πολλέ δυνατότητε, αλλά πρέπει κάπω να τι εκμεταλλευτούμε και πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι συνέπειε. Καταρχά πρέπει να ενισχύσει την δέσμευση και των πακιστανικών αρχών για καταπολέμηση τη τρομοκρατία. Δεν έχει νόημα να μπούμε σε μια ανάλυση εις βάθος για να ξέρουμε για παράδειγμα αν ε, η ήταν ε, ανικανότητα ε, η συνενοχή των πακιστανικών αρχών. Νομίζω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή της κατάστασης αυτής της δύσκολης για να πιέσουμε ακόμη περισσότερο και να ζητήσουμε από τους Πακιστανούς να, ε, ε, να συνεργαστούν περισσότερο μαζί μας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, δεν ξέρω κατά πόσο τι ακριβώς συνέβη στο Πακιστάν, αλλά εδώ και κάποια χρόνια ε, ο Πακιστανικός ε, ε, στρατός και συχνά και οι στρατιωτικές δυνάμεις στο Πακιστάν είναι πολύ συχνά θύμα οι ίδιοι τρομοκρατικών πράξεων. Και τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και στο Αφγανιστάν και ελπίζω να ε, μπορέσουν οι Ταλιμπάν να αποστασιοποιηθούν από τον Αλκάιντα και να συμμετέχουν περισσότερο στην ε, διαδικασία συμφιλίωσης. Τρίτο σημείο, με τεράστιο ερωτηματικό βέβαια, είναι το να ξέρουμε κατά πόσο μετά από 10 χρόνια ε, που είχε δημιουργηθεί έτσι μια απόγνωση από πλευράς ε, ε, αμερικανικού πληθυσμού, ο θάνατος του Οσάμα Μπιλάντεν θα μπορούσε να δημιουργήσει μια καλύτερη διάθεση από πλευράς προς το, για το Κογκρέσο, για παράδειγμα, σε σχέση με το όλο θέμα ε, για παράδειγμα, ε, είδαμε ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ήθελε να περάσει μια προσέγγιση πιο ε, ευρα, ευρωπαϊκή και να αφήσει αυτόν τον παγκόσμιο πόλεμο κατά της τροποκρατίας, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τον προκάτοχο του. Δηλαδή, ήθελε να δικαστούν ορισμένοι σε ποινικά δικαστήρια κανονικά. Ε, δεν προσπάθησε να δεν μπορούσε να κάνει όλα αυτά όσο είχε πει, όσα είχε πει για παράδειγμα το πλήρες κλείσιμο του Γαντανάμου, κατάφερε να κάνει περίπου το 50%, είναι πάρα πολύ δύσκολο, ε, το, ε, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, βέβαια πήρε πολύ σοβαρές αποφάσεις όσον αφορά τα, την ε, έκδοση ή όσον αφορά τα βασανιστήρια. Υπάρχει λοιπόν παν, παράλληλα μια τεράστια συζήτηση αρκετά έντονη στις ΗΠΑ σε σχέση με την πολιτική του Ομπάμα και ελπίζω να μπορέσει ο κύριος Ομπάμα να ολοκληρώσει τους στόχους που είχε εξαγγείλει. Πρέπει όμως να πούμε ότι παρά τους θετικούς στόχους, ο, θανάτο, ο θάνατος του Οσάμα Μπιν δεν σημαίνει το τέλος της ε, Αλκάιντα, ούτε το τέλος της τρομοκρατίας, δυστυχώς. Πολλές φορές είχα την ευκαιρία να πω και ίσως είναι κάπως απλοϊκό να παρουσιάζεται έτσι η απειλή, όλο και περισσότερο περίπλοκη και πιο διαφοροποιημένη είναι η απειλή και συνεπώς είναι πολύ πιο δύσκολο να την εντοπίσουμε, τουλάχιστον με τα μέσα ε, μυστικών πληροφοριών που έχουμε. Ε, Έχουμε συγκεκριμένες ε, οργανώσεις ε, που είναι πολύ ε, δραστήριες στην περιοχή τους και καμιά φορά βγαίνουν από την δική τους περιοχή και δραστηριοποιούνται Εκτός, για παράδειγμα, πούμε, βλέπουμε τι γίνεται στην Ιεμένη, η Αλκάιντα στο Ισλαμικό ε, Μαγκρέπ, η οποία εξακολουθεί να στρατεύει κόσμο και ε, ήταν ε, προφανώς αποσυνδεδεμένη από το πυρήνα ε, της Αλκάιντα στο Πακιστάν. Η Αλκάιντα στο Ιράκ δεν έχει εξαφανιστεί και φυσικά δεν αναφέρομαι γιατί ε, υπάρχει η Ελσαμπάπ στη Σομαλία, δεν είναι όμως ακριβές παρακλάδι αυτό της, ε, της Αλκάιντα, είναι όμως αρκετά συνδεδεμένη και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να την αναφέρουμε. Και στο Τατζικιστάν υπάρχει, ε, υπάρχουν κάποια, ε, ε, κάποιες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται από το Βόρειο Κάφκασο προς την Ασία. Οι foreign fighters λοιπόν όπως τους λέμε, οι ξένοι αγωνιστές που ζουν στην Ευρώπη, και που θα πάνε στα διάφορα hot spots ε, να ε, εκπαιδευτούν και ενδεχομένως να αναλάβουν επιθέσεις εναντίον των δικών μας κρατών. Για παράδειγμα στο Ντίσελντορφ με τι έγιναν συλλήψεις ε, ακόμη και Πακιστανών και η Γαλλία μάλιστα συνέλαβε ορισμένους νέους που συμμετείχαν στις ε, στην, ε, στις, στις οργανώσεις αυτές. Γύρω στα 20-30 άτομα γαλλικής υπηκοότητας ε, θα έπρεπε να υπάρχουν κανονικά στη συγκεκριμένη οργάνωση, όμως αναφέρονται επίσης και άλλα νούμερα, όπως 200 Γερμανοί για παράδειγμα στην Αυγανοπακιστανική ζώνη και κάποιοι μάλιστα καμιά εβδομηταριά είχαν επιστρέψει και στη Γερμανία. Δεν είναι τεράστια τα νούμερα, αλλά έχουν κάποια σημασία τα νούμερα αυτά. Και κάτι δεν είναι τεράστια λοιπόν τα νούμερα όπως σας ε, είπα και σας είπα μόλις, ε, απλώς υπάρχουν πάρα πολλοί σύνδεσμοι είτε με τον κεντρικό πυρήνα της Αλκάιντα είτε με παρακλάδια της ε, Αλκάιντα ε, που έχουν την τάση ριζοσπαστικοποίηση όλο και περισσότερο. Η Εμένη, για παράδειγμα, όλο και ενθαρρύνει περισσότερο με εντελώς τυχαίο τρόπο ε, κόσμο να κάνει επιθέσεις, ακόμη και αν δεν είναι οργανωμένες οι επιθέσεις αυτές. Το Μαρακές, κατά τη γνώμη μου, από ό,τι κατάλαβα τουλάχιστον από τις πληροφορίες που έλαβα, ε, ήταν αποτέλεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας... Ε, ε, είδαμε επίσης τι συνέβη και σε άλλες ε, περιοχές, όπως για παράδειγμα στη Λιέγη, ε, ένας τσετσένο ο οποίος συνδέθηκε με την όλη διαδικασία των σκίτσων του Μωάμεθ. Είναι γεγονός ε, ότι υπάρχουν ε, περιοδικά όπως για παράδειγμα το Inspire ε, που είναι ένα από τα βασικά περιοδικά, από τα σημαντικά περιοδικά στις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι πάρα πολύ καλοφτιαγμένο και καλοί νέους όσο το δυνατόν περισσότερο να χτυπούν όποτε μπορούν να χτυπήσουν. Οπότε λοιπόν το συμπέρασμα των Υπουργών ήταν να ε, πούν ότι υπήρξαν συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στι Ηνωμένε Πολιτείε μετά από το θάνατο του Μπιν Λάντεν και αυτό συμπληρώνεται, εντάξει δεν έχω πολύ συγκεκριμένε ε, πληροφορίε, αλλά δεν θέλει και πολύ για να το καταλάβουμε, είναι προσπάθειες να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενα αντίπεινα στο άμεσο μέλλον. Έχουμε ε, σύντομα το Σεπτέμβριο τη δέκατη επέτειο των δρομοκρατικών επιθέσεων στι ΗΠΑ και γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Αυτά λοιπόν για το θάνατο τώρα του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Για την Αραβική Άνοιξη τώρα να πω ορισμένα πράγματα. Ε, δεν έχω να σας πω τίποτε πολύ πρωτότυπο, αλλά είναι γεγονός ότι είναι πραγματικά κάτι το πολύ αισιόδοξο σε σχέση με όλη αυτήν την ε, ζωφερή ρητορική του Οσάμα Μπιν Λάντεν πάρα πολλά χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ε, μια μη βίαιη ε, προσπάθεια ετήματος σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας ε, μέσω πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα βέβαια και αυτό είναι εξαιρετικά νέα ότι μπορεί να υπάρξει δημοκρατία που θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης, που θα δώσει τη δυνατότητα σε αντιφρονούντες να εισακούονται ε, και θα οδηγήσει και σε κράτος δικαίου. Είναι νομίζω η καλύτερη λύση για να μπορέσουμε να προλα... να προλάβουμε και να μειώσουμε την τρομοκρατία. Κάτι το οποίο εμένα με απασχολεί βέβαια είναι ότι πολλές από αυτές τις χώρες, ε, για παράδειγμα Αίγυπτος και την Ισία, για πολλούς λόγους ε, από, ε, δυναμώνουν τα, τις ε, μυστικές τους υπηρεσίες για την ώρα, ε, απελευθερώνουν πολιτικούς κρατούμενους από τις φυλακές τους, αλλά μεταξύ αυτών υπάρχουν και κάποιοι που ε, επιδίδονται στο τζιχάντ και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, και υπάρχει βέβαια και το θέμα στη Λιβύη, γιατί στη Λιβύη υπάρχει όλο και περισσότερος ε, εξοπλισμός και αν, υπάρξει και αν συγκεντρωθεί σε λάθος χέρια και στη Λιβύη και στην Ιεμένη έχουμε φιλετικές δομές ουσιαστικά και επομένως μπορεί να αποτελέσουν ε, κέντρα τρομοκρατικής δράσης, κέντρα τζιχάντ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε την ε, απάντησή μας σε μεγάλο βαθμό, την στρατηγική μας. Πρόκειται για μια στρατηγική που εγκρίναμε το 2005. Πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής ε, και συνεκτικοί. Εγώ επιμένω πάρα πολύ στην πρόληψη και χαίρομαι ιδιαίτερα ότι που είδα ότι η Επίτροπος ε, Μάλμστρομ, αρμόδια για την εσωτερική ασφάλεια, ε, έδωσε συγκεκριμένα μέτρα ε, προς ε, από το Συμβούλιο βάσει δύο αξώνων και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και καλό θα ήταν να την υποστηρίξουμε. Ένα ακόμη πολύ μεγάλο θέμα, δεύτερο μεγάλο θέμα το οποίο δημιουργεί πολλές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και καταλαβαίνουμε γιατί, είναι τα νέα μέσα συλλογής δεδομένων που προτείνει το Συμβούλιο, που θα ήθελε το Συμβούλιο, όχι από τους δικαστές και από την αστυνομία, αλλά από ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηλαδή τηλεπικοινωνίας, προμηθευτές ίντερνετ, αεροπορικές εταιρείε, το PNR για παράδειγμα, ε, ή για παράδειγμα το SWIFT που έδωσε σημαντικές πληροφορίες για θέματα χρηματοδότησης ε, θα υπάρξει λοιπόν μια πρόταση μετά το καλοκαίρι ε, ενώ ένα σύστημα TFTP, Terrorist Financing Tracking Program, το οποίο βέβαια ε, προκαλεί πάρα πολλές συζητήσεις Εγώ δεν λέω βέβαια ότι θα πρέπει να υπάρχει ελευθερία και δικαιοσύνη, απλώ πιστεύω ότι χρειάζονται πιο πολλά προσωπικά δεδομένα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, γιατί είναι πολύ πιο περίπλοκη η απειλή και είναι πολύ πιο δύσκολο για τι ε, χώρε μα να αντιμετωπίσουν ύποπτε τρομοκρατικέ οργανώσει ή, εν περιπτώσει, ύποπτε τηλεφωνικέ κλήσει κλπ. Πρέπει να είμαστε πραγματικά πολύ πιο στεναροί στην προσπάθειά μα και νομίζω ότι εκεί πρέπει να πέσει το βάρο. Υπάρχει ένα ακόμη τρίτο κομμάτι, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι αυτό που μάθαμε μετά τις ε, ε, επιθέσεις στην Ιεμένη. Ε, για παράδειγμα, δύο πακέτα με εκτυπωτές που είχαν εκρηκτικά μέσα και θα Ε, ε, για τη διάρκεια των πτήσεων. Είναι κάτι το πολύ φιλόδοξο. Πρέπει να δούμε και εμείς πώς θα αλλάξουμε αναλόγως την ε, νοοτροπία μας. Δηλαδή πρέπει και σε εθνικό ε, επίπεδο, και δεν είναι όλα τα κράτη-μέλη ικανά να το κάνουν αυτό, είναι συντονισμός τελωνίων, αεροπορικών ε, εταιριών και όλων των τομέων των μεταφορών, ακόμα και το DHL για παράδειγμα. Πολλές φορές δραστηριοποιείται στον κόσμο σε τέτοιο μεγάλο βαθμό που θα μπορούσε να μας ε, βοηθήσει. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο για μια τέτοια εταιρεία να εξασφαλίσει την ασφάλειά της αν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε συγκεκριμένα ευαίσθητα δεδομένα που προέρχονται από μυστικές υπηρεσίες. Όμως υπάρχουν κάποια προβλήματα ρευστότητα μεταξύ ε, πληροφοριών που ε, πηγαίνουν από το δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα κλπ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρώτη φορά προσπαθεί να αναπτύξει ε, ανάλυση κινδύνου βάσει των δεδομένων που λαμβάνει από τα κράτη-μέλη και μάλιστα σε διάλογο με τους διάφορους κλάδους προσπαθεί να δει τις πιθανότητες και τον αντίκτυπο μιας επίθεσης και επομένως προσπαθούμε έτσι να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις όταν κάτι όταν κάποιος ε, ε, ε, υψηλού κινδύνου, για παράδειγμα από τη Μαυριτανία, ε, ε, κυκλοφορεί με κάποια από τα μέσα μεταφοράς. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Να δούμε λοιπόν αυτά που λέτε για το Πακιστάν. Ε, παρακαλώ υποστηρίξτε μέσω του προπλογισμού το θέμα αυτό και ε, την αστυνομία και το δικαστικό σώμα του Πακιστάν το βοηθούμε για καλύτερη λειτουργία για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας 15 εκατομμύρια ευρώ χαμηλό ποσό σε σχέση με αυτά που προσφέρουν στο Πακιστάν Αμερικανοί χρειάζεται επαγγελματικός χαρακτήρας στην αστυνομία και στο δικαστικό σώμα και η προσέγγιση είναι στρατιωτική μόνο δυστυχώς και οι ε, πλευρές δικαστικής δεν μπορούν να κυνηγήσουν όπως πρέπει τους τρομοκράτες, δεν μπορούν να έχουν αποδεικτικά στοιχεία και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται αυτή τη αδυναμία του Πακιστών να κρίνει τους ε, όσους ε, ε, έκανε αυτή την απόπειρα στη Βομβάη και ακόμη κάτι το να κρίνει κανείς τρομοκράτες σε μια ποινική δίκη καλό θα ήταν ταυτόχρονα και για τη δικαιοσύνη αλλά και το καλύτερο μήνυμα για τους τρομοκράτες ε, ότι είμαστε δυνατοί και ότι είναι απλοί ε, εγκληματίε και όχι υπέρ μιας ε, κάποιας ιδέας. Ακόμα κάτι, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει το Κοινοβούλιο είναι ότι νομίζω ακριβώς γρήγορα θα πρέπει να υπάρξει ένας μηχανισμός για να βοηθήσουμε τις χώρες σε μεταβατική περίοδο δημοκρατίας όπως την Αίγυπτο και την Τουνησία πάνω απ' όλα και να μπορέσουν να επαναδιαρθρώσουν ε, θέματα ασφάλειας ε, και με κατάλληλες υπηρεσίες, αλλά να σέβονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό που κάναμε μετά από την πτώση του τείχους του Βερολίνου με ένα σύστημα, αυτά τα twinnings, ε, σύζευξη και οι δικοί μας, οι μυστικές υπηρεσίες στη Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο κλπ. βοήθησαν τους συναδέλφους εκεί να έχουν ε, υπηρεσίες που να είναι αποτελεσματικές ε, και όπως τις τάζεις, τις εκοριτάτε κλπ. Τουρκική Γερμανία, Ρουμανία, το ένα άλλο και χρειάστηκε ακριβώς να διορθεί αλλά δεν μπορούμε έτσι να, μην έχουμε, να έχουμε ένα κενό ασφάλειας και η πρώτη απάντηση ήταν πολύ καλή από την κυρία Άστον και από την Επιτροπή στα γεγονότα αυτά στις 11 Μαρτίου στο Συμβούλιο εκεί ήταν κάτι πολύ πολύ το καλό σχετικά με την οικονομική υποστήριξη στην νεολαία, στην ε, εσωτερική μετανάστευση. Όλα αυτά και ταυτόχρονα θα πρέπει να αναφέρουμε και την ασφάλεια γενικά, είτε με αυτή το του είναι τη σύζευξη, είτε το CSDP, αυτή τη μεταρρύθμιση σε θέματα ασφάλειας ε, από συναδέλφια ακριβώς στην υπηρεσία, κάνουν τις απαραίτητες αναλύσεις και θα πρέπει να επιμείνουμε και αυτή τη στιγμή την Ισία δεν μας έχει ζητήσει τίποτα μέχρι τώρα αλλά χρειάζονται αρκετά χρήματα και θα δείξω μια κάποια λογική και να ε, μπορέσουμε ταυτόχρονα να πούμε και εμείς ε, δεν είναι μόνο το more for more και ταυτόχρονα θα πρέπει να συνδυάσουμε τη βοήθειά μας με ορισμένα πράγματα που μας ζητούνται σε θέματα ασφαλείας. Τέταρτο στοιχείο, η επικοινωνία, κάτι που με έκανε εντύπωση όχι μόνο εμένα μετά από το θάνατο του Μπεν Λάντεν για τα κράτη-μέλη και οι διάφορα ε, θεσμικά όργανα στις Βρυξέλλες πώς αντέδρασαν και εγώ ίδιος, εγώ συνέταξα το ανακοινωθέν μου που δεν ήταν όμως όλα αυτά με συντονισμένο τρόπο. Καλό θα ήταν λοιπόν στα πλαίσια της δεκάτης επαιτίου μετά από τα γεγονότα της, ε, στη Νέα Υόρκη θα πρέπει να μπορέσουμε να περάσουμε ένα μήνυμα που να συγκλίνει με τα υπόλοιπα. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο σημείο. Τώρα για τα υπόλοιπα. Το καλό το νέο ποιο είναι. Το Συμβούλιο Περγών Εξωτερικών ε, υιοθέτησε τις 21 Μαρτίου μια σχετική στρατηγική που είχα ξεκινήσει εγώ πριν από 2,5 με 3 χρόνια και προσπαθούσα με το συνάδελφα για την ανάπτυξη να δούμε κάπου ακριβώς που θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα πείραμα έτσι χωρίς ε, ιδεολογικά προηγούμενα μια προσέγγιση ολοκληρωμένη και ε, συγκλίνουσα ανάμεσα ανάπτυξη και ασφάλεια και αφού είδαμε, επισκεφθήκαμε αρκετέ φορέ επί τόπου τα μέρη αυτά. Νομίζω ότι η στατική αυτή, όπως χαράθηκε, είναι πολύ καλή και με τους συναδελφού από τους για θέματα Ακριβώ παρόμοια και ακριβώ το θέμα τη ασφάλεια είναι κάτι που υποστηρίζουν και 27 υπουργοί εσωτερικών όχι μόνο από τη Γαλλία, την Ισπανία και του άμεσου γείτονε. αλλά και 27 θέλουν να αφιερώσουν μέσα και μάλιστα σημαντικά υψηλά οικονομικά και ανθρώπινου προσωπικού για θέματα παρόμοια ασφάλεια και ανάπτυξη και για να επανέλθουμε στο θέμα ακριβώ αυτό οι Τουαρέγ, οι μισθοφόροι που επεστρέφουν στα βόρεια του Μαλή και στην ε, Νιγέρα. Εδώ είναι ιδιαίτερα σχέδια για να δείξουμε ακριβώς τον πληθυσμό του βορρά του Μαλή ότι αλλάζουν τα πράγματα έτσι. Αυτό για να ενισχύσουμε όλα αυτά, στην ασφάλεια, διπλωματικά κλπ. Πολλά θα πρέπει να γίνουν και για την πρόληψη επίση για να μην υπάρξει ένα ριζοσπαστικός νέο χαρακτήρα. αυτό στον Ήγηρα και λιγότερο ε, στη Μαλή και πολύ στη Μαυριτανία. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται για να έχουμε τα μέσα για να προλάβουμε την εξέλιξη προ ένα ριζοσπαστικό Ισλάμ. Και υπάρχουν διάφορε πρωτοβουλίε που αναλαμβάνονται στην περιοχή εκείνη. Χαίρομαι η Υπουργή Εξωτερικών του Μαλή, Μαϊγκά, ο νέο υπουργό, ο οποίο με την ε, Νίγηρα, τη Μαυριτανία και την Αλγερία συναντήθηκαν ε, με, συναντήθηκε με του ομολόγου του τη Βλαμπαμπέζα και προσπάθησε να επιταχύνει την όλη κατάσταση γιατί ε, με την Αλγερία κάτι το καινούριο επίση, ένα γενικό α πούμε έτσι επιτελείο με κοινέ συγκλίνωσε θέσει και σύμφωνα με τον τύπο και Σμύρνη το φθινόπωρο ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση στι ΗΠΑ. Θα λάβει χώρα, θα οργανιστεί στην Αλγερία μια σύνδεση και μια συνάντηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και με τον Καναδά, τι ΗΠΑ, την Ιαπωνία, την Αυστραλία θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε για την πρόθεση αυτή τη στρατηγική. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Και ακόμη κάτι, ένα από τα σημεία τα οποία είπατε και εσείς ο ίδιος. Για να δούμε πώς ε, το νέο πλαίσιο, η νέα αρχιτεκτονική δεσμική λειτουργεί μετά από τη συνδική της Υπάρχουν ε, νέοι που μετέχουν ε, και όλα αυτά προχωρούν βέβαια η υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων και όλα αυτά είναι αρκετά λογικά για να μπορέσουμε να δούμε τη νέα θέση των διαφόρων εταίρων. Αυτή είναι η υπηρεσία λοιπόν και το Συμβούλιο και να σας πω επίσης ότι σύμφωνα με λέγω αποτελώ εγώ και εγώ ένα θεσμό, όχι για τις αρμοδιότητες λοιπόν, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί κανείς να βοηθήσει για καλύτερο συντονισμό ευρύτερο ανάμεσα σε όλα αυτά που γίνονται από τους μεν και του δε. Αυτό δεν είναι απλά. Το κάθε κράτος μέλος ε, καταλαβαίνει τη δυσκολία για να μπορέσουν οι διπλωμάτες, υπεύθυνοι από το Υπουργείο Εσωτερικών και υπεύθυνοι από τις υπηρεσίες πληροφοριών, πώς, θα μπορούν να συνεργαστούν μαζί, μαζί και η Επιτροπή έχει σημαντικά με και αυτή ακριβώς εξωτερική ασφάλεια έχει ιδιαίτερη σημασία και ο Άλστρομ ε, δείχνει, παίζει ιδιαίτερα ενεργό ρόλο και τώρα τελευταία ας πούμε για τα ναρκωτικά σε μια ενδιαφέρουσα ε, διάλεξη στην Πορτογαλία και όλα αυτά να χαρακτηρίζονται από ένα λογικό κοινοπλαίσιο και επίσης η κόψη και η κοζή η νέα επιτροπή ε, μέσω της Σύνθηκης της Σαββόνας ε, από την 1η Ιουνίου θα έχουμε μια πρώτη συνάντηση, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, για να δει κανεί με ποιο τρόπο θα μπορέσει να εργαστεί καλύτερα, να συνδυαστούν αυτοί οι δύο κόσμοι και αυτό μπορούμε να κάνουμε ξεκινώντας ανάμεσα στην PSDC και στην αποστολή αυτή και στα μέσα, τα εργαλεία που έχουμε ε, μέσω της ε, δικαιοσύνης και των συνολικών υποθέσεων, η Europol, η Eurojust, Sepol, Frontex, ε, όλα αυτοί και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και αυτό με απασχολεί ιδιαίτερα αρκετές φορές υπέβαλα, ερωτήσεις, υπέβαλα προτάσεις στις αντιπροσωπείες για θέματα ακριβώ και στρατιωτική ασφάλεια και εσωτερική ασφάλεια και ορισμένοι έχουν ακριβώς τις πρεσβείες τους ε, άτομα που ασχολούνται με αυτό και στην Αλγερία δεν ξέρω ότι δεν νομίζω δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πληροφορίες τόπου αν δεν υπάρχει κάποιος που να έλθει σε επαφή στενή με τους υπεύθυνου. κάτι λοιπόν που θα πρέπει όσο γίνεται πιο γρήγορα να εξελίξουμε και ακόμη κάτι στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων 10 Ιουνίου θα οργανωθεί αυτό και που θα ε, καταλήξουν σε συμπεράσματα το πώς θα βελτιώσουμε ακόμα καλύτερα χρήση αυτών των εργαλείων ώστε ακριβώς να λεφθούν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία για την ε, εσωτερική ασφάλεια από όλου. Κάτι ακόμα αποτελεί ευχή των Υπουργών Εσωτερικών, η κυρία Άστον και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να μπορέσουν να οργανωθούν κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ανάγκες γιατί αν δεν γίνει εκεί, έτσι πρέπει να γίνει κάπου εδώ πέρα από το ε, ε, και τα αεροπλάνα μεταφορών ας πούμε για εμπορεύματα που θα πρέπει να οργανωθούν και λόγω της διασπόρας αρκετοί από τους Ομαλούς ζουν σε μέσα και στη Σκανδιναβία που θα πρέπει να φτάσουν στην και θα πρέπει να μπορέσουμε να τα συνδυάσουμε όλα αυτά, να τα οργανώσουμε καλά και επίσης ένα συντονισμό των οικονομικών μέσων, κάτι που προσπαθώ να κάνω εγώ και οι υπηρεσίες και δράσεις ε, με άμεση ε, πρόσβαση στα μέσα σταθερότητος και ξέρετε ότι πρόκειται για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, για τη στήριξη ε, καλής γειτονίας κλπ. και όλα αυτά που θα μπορούσαν ε, να βοηθήσουν ε, στην εσωτερική ασφάλεια. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε σίγουροι ότι συνεργαζόμαστε γίνεται καλύτερα με το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα να μην έχουμε είτε μία επέμβαση είτε πολλαπλή επέμβαση. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για αυτά που είπατε κύριε Πρόεδρε. και παραμένω σε ορισμένα θέματα τα οποία καλά κάνατε και υπενθυμίσατε διότι δεν είχαμε υπενθυμίσει επαρκώς στην επιχείρηση του του Ομπάμα εναντίον του Μπεν Λάντεν ότι τα θύματα ήταν ιδίω μουσουλμάνοι και είναι ένα θέμα το οποίο δεν τονίσαμε επαρκώς στις παιδαγωγικές προσπάθειες που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει κανείς να επιλύσει αυτό το, αυτή την εγκληματική πτυχή είτε πρόκειται για το Ιράκ, για το Πακιστάν, για το Αφγανιστάν όπου τα θύματα είναι μουσουλμάνοι. Το δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να τονίσω είναι η Αλκάιντα στη, στο Ισλαμικό Μαγκρέμπ και ε, έχουμε συζητήσει επανειλημμένως αυτή την πρόκληση η οποία όντως απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη με διάφορες μορφές, με δυνατότητες που αυξάνονται και γι' αυτό η κρίση στην ε, Ευρώπη δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Αναφέρατε τους μισθοφόρους, ε, την διακίνηση ε, όπλων και η κατάσταση στη Λιβύη μπορεί να επιδεινώσει την επέκταση αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων στο Μαλί, στο Νίγηρα και στην Μαυριτανία. Και θα θίξουμε το θέμα αυτό στη συνέχεια. Βεβαίως αντελήφθην αυτό που είπατε για το Πακιστάν και στην δικαστική αρρωγή στο Πακιστάν διότι πρέπει να επικεντρωθούμε επίσης και εις το δικαστικό εμπόδιο για την τρομοκρατία και όχι μόνο τις άλλες ε, εκδοχές όπου θα πρέπει επίσης να βοηθήσουμε την αστυνομική και δικαστική αρρωγή. Αναφερθήκατε σε risk assessment, αξιολόγηση του κινδύνου, αλλά αυτή γίνεται από την Επιτροπή, όντως αυτό είναι το πρόγραμμά μας από την αρμόδια Γενική Διεύθυνση στην Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει του άρθρου 4 Έχουμε τις, ε, την πληροφόρηση εκτός του θεσμικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για να συντονίζουμε στρατηγικά δεδομένα αναλόγως των καταστάσεων. Αλλά ε, δεν εφαρμόζεται ακόμη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Πρέπει λοιπόν να διαστραβρώσουμε τις, ε, την πληροφόρηση για την αντιτρομοκρατική για τρομοκρατική Απειλεί με τους κινδύνους στα αεροδρόμια, στους χώρους, στις χώρες, Μαυριτανία κτλ. Και αναλόγως να αξιολογήσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσουμε εάν θα ελέγξουμε τα φορτία παραδείγματος χάρη αναλόγως του κινδύνου και του πόσο ευάλωτοι είμαστε. Είναι κάτι που θα πρέπει να μπορέσουμε να επεκτείνουμε και σε άλλους τομείς τα φορτία π.χ. είναι ένας τομέας τέτοιος. Η Άννα Γκόμες, ε, παρακαλώ να μας πείτε κάτι για αυτή τη μετακίνηση στη Λιβύη και την διασύνδεση με τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Πέρασα μία εβδομάδα στη Βενγάζη και πέρασα από όλε τι ζώνε που ήταν ελεύθερε, μεταξύ των οποίων και το Frontline. Και συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπατε, ότι πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να να αποστείλει ε, μία, να αναπτύξει μία αποστολή ε, πά, για να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. Και παράλληλα θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχω ότι δεν έχω καμία απόδειξη ε, διείσδυσης τρομοκρατικών οργανώσεων ε, στις περιοχές στις οποίες κυκλοφόρησα εγώ. Είναι άνθρωποι, για παράδειγμα γιατροί, που έχουν εν πάση περιπτώσει τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή τους ε, για να απελευθερώσουν τη χώρα τους. Μάλιστα ήρθαν νέοι να με δουν για να μου πούνε πώς αισθάνεται ένας μουσουλμάνος προσβεβλημένος από το γεγονός ότι τους θεωρούσαν ε, ως, ε, τους θεωρούσαν τρομοκράτες και μάλιστα κάποιος ε, ε, μου είπε συγκεκριμένα ότι ως πραγματικός μουσουλμάνος με, με, με, με λυπεί, με πονά πραγματικά το γεγονός ότι μας θεωρούν αυτομάτως τρομοκράτες. Και πρέπει να πω και ως Ευρωπαία γυναίκα δεν, είχα κανένα πρόβλημα, δεν είχα κανένα πρόβλημα ε, στις ε, σχέσεις μου, ούτε είδα ιδιαίτερα ε, φονταμενταλιστική προσέγγιση τέλος πάντων προς εμένα. Στις υπόλοιπες περιοχές της Λιβύης ε, υπάρχει αναγνώριση ότι αν συνεχιστεί η ε, σύγκρουση δίνει τη δυνατότητα διείσδυσης τρομοκρατικής ε, και από, την, από τα νότια σύνορα, τα οποία ελέγχονται πολύ λίγο και αυτό πραγματικά δημιουργεί ανάγκη εποπτεία στα σύνορα, ενίσχυσης του εμπάργου όπλων και προσπάθειες εξέτασης τέλος πάντων της ε, διείσδυσης των μισθοφόρων. Ε, ξέρουμε πολύ καλά την, ε, τι κάνει σχετικά με αυτό το θέμα αυτό. Από την Αλγερία κιόλα φέρνει μισθοφόρους ο, ο Καντάφη. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια αποστολή εκεί και συμφωνώ απόλυτα με την επίσκεψη της κυρίας Άστον και με την ύπαρξη ενός γραφείου εκεί και υποθέτω και ο ίδιος ο κύριος Δεκέρκοφ θα μπορούσε να μεταβεί. Είναι πάρα πολύ σημαντική όλη αυτή η προσπάθεια και για τους νέους που βρίσκονται ε, στα ε, φυλάκια, στα σύνορα. Ε, για παράδειγμα, ένας Γάλλος πολίτης έχασε τη ζωή του προσφάτως και μου το εξήγησαν ότι απλώς ένα checkpoint κάποιοι νέοι που είχαν περάσει, εν πάση περιπτώσει, μια στρατιωτική εκπαίδευση ήθελαν κάπως να επιδείξουν, εν πάση περιπτώσει, τις ε, ε, ε ιδιότητες που μόλις είχαν αποκτήσει και, εν πάση περιπτώσει, κάπως έτσι έγινε και έχασε τη ζωή του ο Γάλλος πολίτης. Ε, δεν ήταν ακριβώς τρομοκρατική επίθεση, οπότε θα ήθελα να σας ζητήσω, ε, κύριε Ντεκέρχοπ, να επιμείνετε για αυτή την αποστολή. Η κυρία Άστον είχε εξαγγείλει κάτι τέτοιο, αλλά δεν έγινε τίποτε. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για να υπάρξει μια τέτοιου είδους αποστολή για την ε, στο πλαίσιο της EU4 ε, ε, Λιβύη. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Και ένα ερώτημα θα ήθελα να σας θέσω. Συμφωνώ και εγώ απολύτως με όλα αυτά που είπατε στο τι πρέπει να ζητήσουμε από τις γειτονικές χώρες, όπως για παράδειγμα την Ισία. Αναφερθήκατε όμως στο Σαχέλ. Το Σαχέλ καταλαβαίνει... για παράδειγμα, η Γκουινέα Βυσάου καταλαβαίνει ε, το πρόβλημα και τη σχέση που έχει με το πρόβλημα, για παράδειγμα η εγκληματικότητα που υπάρχει για το λαθεμπόριο ναρκωτικών, για παράδειγμα πάρα πολύ γρήγορα υποστηρίζει την ε, ε, οργανωμένη τρομοκρατία και την πειρατεία. Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω και κάτι ακόμη για το Πακιστάν. Συμφωνώ απολύτως με την προσπάθεια αυτή που προτείνεται και θα έπρεπε να σας υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απλώς αναρωτιέμαι αν δεν αντιμετωπιστεί το ζήτημα του Κασμίρ, που είναι πραγματικά το κίνητρο του Πακιστάν και του Πακιστανικού στρατού, δεν πρόκειται πουθενά να καταλήξουμε. Δεν θα καταφέρουμε πολλά και μιλάμε για μια χώρα που έχει πυρηνικά όπλα που θα μπορούσαν να πέσουν σε λάθος χέρια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη προτεραιότητα. Ευχαριστώ. Euh, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κερκόφ ε, για τα όσα μας είπε. Επιτρέψτε μου να πω να αφιερώσω τα 30 πρώτα δευτερόλεπτα στον πρόεδρο της μας ε, για να ζητήσω για, συγγνώμη για την απουσία μου για το σημείο 4. Είμαι σκιώδης συγητής. Ε. Ξέρω ότι ο κ. Πασκού βοήθησε και σύμφωνα με όσα είχε πει η ομάδα μου. Αλλά σχετικά με όσα είπατε εσείς, εγώ παρακολούθησα το θέμα του αγώνα κατά της τρομοκρατίας ε, σε ευρωπαϊκή κλίμακα και κοινοβουλευτική επίσης από την προηγούμενη διευθυντία του Κοινοβουλίου. Τώρα, ίσως επειδή οι πολίτες από χώρες που ιστορικά υποφέραμε από μια σκληρή τρομοκρατία και τώρα και τα τελευταία χρόνια όπως έγινε και το 2004 μια απόπειρα ε, Ισλαμικής προέλευσης. Ε, να σας πω ότι προσέχουμε ιδιαίτερα, ίσως περισσότερο από άλλους, το πρόβλημα αυτό. Ήδη λεκτικά τουλάχιστον είμαστε αντίθετοι με την τότε βορειοαμερικανική άποψη για την πόλεμο κατά ε, Με τον τρόπο αυτό γιατί αυτό προϋπέθεται αναγνώριση και των αντιπάλων και στρατιωτική αντιμετώπιση και υποδαβλίζαμε την Ισλαμοφοβία, έτσι. Η Ευρώπη δεν είχε ακολουθήσει σαν σύνολο ενιαίο την αντίληψη αυτή και η νέα Αμερικανική διοίκηση ούτε επίση τελικά επέλεξε αυτό το τρόπο για τη μάχη κατά της τρομοκρατίας που έχουμε τώρα μια διαφορετική αντίληψη και προσπαθούμε να αντιδράσουμε αποτελεσματικά στα πλαίσια όμως ενός κράτους δικαίου με εγγύσεις και όχι μόνο για ηθικούς λόγους αλλά και για λόγους αποτελεσματικότητας. Αυτό μας διαφοροποιεί ακριβώς ακόμα περισσότερο από τις τρομοκρατικές αυτές ομάδες. Θα ήθελα να εκφράσω την σύμφωνη απόψή μου για όλα αυτά, για την εφαρμογή αυτή. Νομίζω ότι επικεντρώνουμε στην προσοχή μας ε, για την αντιμοκρατία με τον ίδιο τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι είναι μια σημαντική απειλή όλα αυτά. Θα πρέπει να το τονίσουμε, επαναλαμβάνω, γιατί ορισμένοι συνάδελφοι εδώ και ορισμένες ομάδες Κάποιες φορές λένε ότι η αντιτρομοκρατική δράση είναι ουσιαστικά ένα κάλυμα για άλλους στόχους που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με την αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Εντάξει θα πρέπει αν κάτι τέτοιο συμβαίνει να το καταγγέλουμε, αλλά η μάχη κατά της τρομοκρατίας αποτελεί μια μόνιμη ανάγκη. Δεν θα πρέπει να ατονίσουμε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας ε, και μερικές φορές ευτυχώς ευτυχώς ε, για κάποιες περιόδους δεν έχουμε και άσκημα νέα αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να σταματήσουμε τις προσπαθίες μας είναι η τυπική στρατηγική ότι το σημαντικό είναι αυτό που δεν βλέπετε και ε, ότι δεν υπάρχουν νέα και κάτι πρέπει να περιμένουμε προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν και με κατάλληλα εργαλεία για άμεση αντίδραση και στην Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κρατημέλη μεμονωμένα. Έτσι λοιπόν αυτή θα είναι η θέση μας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Ε, βέβαια δέχομαι ε, την, ε, την ε, δικαιολογία και δίνω το λόγο στην κυρία Λόζινγκ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή διότι βλέπουμε και πάλι ότι οι συσχετισμοί είναι πολύ περίπλοκοι γιατί πριν από λίγες ώρες ακούσαμε για τη στρατηγική ε, της καταπολέμησης της ορμοκρατίας και μιλήσαμε για τη διασύνδεση φτώχειας και τρομοκρατίας και ο κύριος Γκάλερ είπε ότι εδώ θα έπρεπε να βασιστούμε περισσότερο στο στρατιωτικό στοιχείο, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ σωστό. Όλα αυτά θα πρέπει να συνδυαστούν και να εξεταστούν από κοινού και ιδίω σχετικά με το Μαγκρέμπ και ε, στο Σαχέλ ο συνδυασμός φτώχειας και Αλκάιντα είναι σαφής. Βέβαια, τίθεται το ερώτημα. Τι ρόλο παίζουν οι, οι ε, στρατιωτικές δαπάνες σε σχέση με τη φτώχεια. δηλαδή ε, τι γίνεται ε, διότι παραμένει, ε, παραμένουν λιγότερα χρήματα για την καταπολέμηση της φτώχειας και να δούμε πώς κατανέμεται αυτό στο Σαχέλ δηλαδή πόσα χρήματα αφιερώνονται στην καταπολέμηση της φτώχειας και πόσα σε άλλους τομείς όπως τη βελτίωση της ασφαλείας. Και θέλω τώρα να επανέλθω σε ένα βασικό θέμα σχετικά με το μαλλί. Στην τελευταία επαφή μου με την Αφρική είχαμε ε, συζητήσει για την κατάσταση στο Μαλί που ήταν ένα πολύ γενικό θέμα και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα υπάρξει επεξεργασία ουρανίου ε, με επιπτώσεις ε, για τον γεωργικό πληθυσμό και δημιουργούν Δε στις ε, διάφορες κινήσεις ε, ε, αντιφρονούντων και πρέπει να ρωτήσω αν σε περίπτωση μέσων που μπορούν να επενδυθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η ασφάλεια μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για να ισχυθεί η πάταξη του πληθυσμού που αντιμετωπίζεται ήδη με στρατιωτικά μέσα. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν κυβερνήσεις ε, οι οποίες θα μπορούσαν να καταπολεμήσουν την τρομοκρατία με τα μέσα που έχουν δεν το πράττουν διότι βρίσκουν ένα τρόπο να ε, επιτύχουν περισσότερη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σχετικά με τον μηχανισμό πάταξης. Δηλαδή ε, μήπως σχετικά με το θέμα της Αλκάιντα δεν δραστηριοποιούνται για να απομυζήσουν περισσότερα χρήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό θέμα που θα έπρεπε να δούμε γιατί θα πρέπει να το εξετάσουμε στο μέλλον. Ένα άλλο συγκεκριμένο ερώτημα σχετικά με την βοήθεια στη βελτίωση του μηχανισμού ασφαλείας συγκεκριμένα στην Αίγυπτο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δραστηριότητες Ευρωπαϊκής Ενώσεως από κοινού με την υπάρχουσα μεταβατική κυβέρνηση για τη βελτίωση του μηχανισμού ασφαλείας και πώς εσείς αξιολογείτε αυτές τις δραστηριότητες ή αν δεν υπάρχουν πώς διαβλέπετε ότι κάτι τέτοιο θα μπορέσει να διαμορφωθεί στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Έχετε το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Για την κυρία Γκόμες, ε, απόλυτα σήμεριζομαι την εκτίμησή σας και σύμφωνα με τις πληροφορίες μου αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει μια διάβρωση, είμαστε 10 και όχι 100. Για τα κράτη-μέλη αυτό που θα ήθελα να επιμείνω και να ενθαρρύνω είναι αυτό το κεντρικό σχετικά με τον Ιούνιο και είχα λάβει το λόγο στην συνάντηση των Υπουργών για αυτό το ίδιο σημείο. Με τον κυρία προσπαθώ επίσης να εκφράσω την απόψη αυτή αλλά στην υπηρεσία εξωτερικών υποθέσεων και με τον νέο υπεύθυνο που συναντήθηκα για τις αποστολές CSDP fact-finding mission ε, που προβλέπονται ακριβώς και ένα συνάδελφο που σήμερα πηγαίνει με αποστολή στο Μαλί για να μπορέσει να εξετάσει το, τα αποτελέσματα θα πρέπει να εξακολουθήσουμε τις προσπάθειές μας, αλλά στις Βρυξέλλες ε, το δέχονται βέβαια αυτό, έχετε δίκιο όμως, ε, γνωρίζετε καλύτερα το θέμα από μένα. Δεν σημειώνεται συνένεση ανάμεσα στα κράτη-μέλη για τη Σαχέλ αυτή καθ' αυτή. Δεν μπόρεσα να πείσω. Αυτό που πιστεύω εγώ είναι ότι αν θέλουμε να βοηθήσουμε και και απαντάω επίσης στην κυρία Λούζινγκ, αυτό που επιθυμούμε καταρχάς να κάνουμε στο Μαλί είναι να χρησιμοποιηθεί το κράτος και να δοθεί μια βοήθεια στο ΠΣΒΕΜ που για να μπορέσει να αποκαταστήσει το κράτος στο Βόρειο Μαλί που είχε εξαφανιστεί και η διαδικασία. Καλή ήταν κατά την απόψή μας ε, γύρω από τη στατική παρουσία να έχουμε και βασικές υπηρεσίες όπως εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές επίσης υπηρεσίες και θα ε, έχουμε προβλέψει 4 εκατομμύρια ευρώ για μια σταθερότητα ακριβώς σε συνεργασία με τις αρχές του Μαλή. αλλά προς στιγμή δεν καταφέραν πίσω όλα τα κράτη-μέλη ότι αυτό που χρειαζόταν απόλυτα ήταν αυτές τις αποστολές να τις χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει γιατί οι αρχές του Μαλή δεν δείχνουν και τόσο αποφασισμένες έτσι να το πω απαλά-απαλά γλυκά-γλυκά εδώ χρειάζεται να βοηθήσουμε και να ενθαρρύνουμε και τις αρχές όλα αυτά να τα προωθήσουν έτσι δραστήρια. Με ένα-δύο συμβούλους στο Μπαμακό, αν πάνε εκεί δεν θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε έτσι. Και εμείς για το θέμα σταθερότητας έχουμε ακριβώς 4,5 εκατομμύρια ευρώ από τη Σιβιπόλ. Είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση με Γάλλους Ισπανούς κλπ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις υπηρεσίες, τις αστυνομικές δυνάμεις για να μπορέσουν να, να διοργανωθούν και εγώ ήμουν εκεί το Νοέμβριο για να ξεκινήσει το πρόγραμμα που είναι πολύ καλό αλλά η κυβέρνηση όμως δεν θα διηθεί έτσι να ξαναγκατασταθεί στο Βόρειο Μαλί. Κάτι χρειάζεται ισχυρότερο, εντονότερο. Θα πρέπει να δούμε τα κράτη-μέλη όπω ακριβώ συμβαίνει με τη Λιβύη ε, και του κινδύνους που ανέφερα. Σω θα πρέπει να δείξουμε περισσότερη αποφασιστικότητα. Τη Γουινέα Μπισάου δεν την καλύπτω ε, Υπάρχει όμω και εκεί μια αποστολή, εντάξει, και σχεδόν έχει ολοκληρωθεί εκεί και θα πρέπει να αποφύγουμε αυτή η κοκαίνη της Νότιας Αμερικής να μην ε, διαβρώσει κι άλλα κράτη όπως στο Βορρά, όπως στη Σενεγάλη κλπ και τους δρόμους στο Σαχέλ και θα πρέπει να δούμε Πώ θα συνδυάσουμε αυτό που κάνουμε σε εσωτερικό και σε εξωτερικό επίπεδο. Ε, συνεργάστηκα με τον ΕΣ ε, για το Σαχέλ σε εξωτερικό επίπεδο, ενώ η άλλη αποστολή ήταν για το δρόμο που ακολουθεί η, ε, το ναρκωτικά με πρωτοβουλία τη Γαλλία και στο Παρίσι μια συνάντηση επίση στην Πορτογαλία, Ηνωμένε Πολιτείε και υπόλοιπο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κατά των δικτύων αυτών με όλα αυτά που κατήγγειλα εγώ. Ίσως θα πρέπει να τα συνδυάσουμε όμω αυτά. Είναι ένα μέρο του έργου στο οποίο ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε τώρα. Συμφωνώ με το Πακιστάν, αυτό που είπατε για το Κασμίρ. Ένα μεγάλο μέρο ε, αυτού του διπλ, αυτής προσπάθειας είναι αυτή η προσέγγιση για να μια μεριά με την Ινδία να δούμε τι γίνεται και από διπλωματικής πλευράς ε, δεν είναι για την κυρία Άστον αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πού βρίσκεται τα κλειδιά, τι θα γίνει, πώς θα τα συνδυάσουμε όλα αυτά, είτε με το Κασμίρ, είτε στο Αφγανιστάν, όλα αυτά και είναι αποτελεί το επίκεντρο τη συζητησή μας με το Πακιστάν. Εσείς, κυρία μου, είπατε για, το Γιάννη. Γιάννης, συγγνώμη. Εδώ θα πρέπει να δούμε τι γίνεται από πολιτικής αστυνομικής πλευράς ε, είναι θέμα και ηθικού και αποτελεσματικότητα ε, Εδώ ε, δεν υπάρχει καμία αναφορά στην καταδίκη της απόπειρας Μαδρίτης. Γιατί, γιατί κρίθηκαν σε μια δίκη ακριβώς δίκη, ορισμένοι απαλλάχθηκαν, ορισμένοι καταδικάστηκαν, είναι φυλακισμένοι και σε αντιμετωπίζουν σαν εγκληματίας. Δεν λέει τίποτα γι' αυτό η αλκαίδα γιατί ακριβώς τους αποκαλούμε ε, εγκληματίας. Ενώ στον Καντάνεμο, α, αυτοί είναι ιδεολόγοι και λοιπά, μαχητές ε, και δίνει έτσι μια λάμψη σε αυτούς μεγαλύτερη και αυτή η διακασία, οι άλλοι που θεωρούνται εγκληματίε, αφαιρεί αυτό το γκλαμούρ, τη λάμψη αυτή από αυτού του εισαγωγικά μαχητέ. Και για τη φτώχεια και την Αλκάιντα, ναι, σε Αλκιντάλ, τι γίνεται από επαγγελματική πλευρά, δεν είναι μόνο μια ομάδα που διακινεί όπλα είτε κοκαίνη. Δίκιο έχετε από τη στιγμή που δεν έχει δυνατότητα να κάνει κάτι το διαφορετικό από οικονομική πλευρά για μια οικονομική ανάπτυξη, δεν θα έχουμε κάτι το θετικό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σα λοιπόν για την ε, οικονομική πτυχή τη βοήθεια Σαχέλ, την ευρωπαϊκή. Ε, εκεί επικεντρώνεται η όλη συζήτηση όχι γιατί ε, χρήματα της ανάπτυξης να πάνε στην ασφάλεια, δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Θέλουμε τη βοήθεια στην ανάπτυξη να τη συγκεντρώσουμε και ακριβώς που υπάρχουν οι απαραίτητοι παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια εξεφάνιση τρομοκρατίας. Και αν δεν μπορέσουμε ε, έξυπνα να κινητοποιήσουμε τα πράγματα, γιατί έτσι σε ε, αγροτικές περιοχές στη μέση της ερήμου δεν μπορούμε να κάνουμε όλα πράγματα υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν φυλές εδώ και εκεί, υπάρχει ξηρασία ε, και εντάξει οικονομική περιοχή λέμε θέμε αλλά ε, περισσότερο εμπόριο είναι στο βορρά του Μαλή με την Αλγερία παρά στην υπόλοιπη Μαλή. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Όπως στην Ευρώπη ίσως διαμεθορικές περιοχές με κινητοποίηση και της Αλγερίας και του Μαλή για να μπορέσουν να συνεργαστούν για το μέρος αυτό λοιπόν. Αλλά η, ε, προσφέρει πάνω από 100 εκατομμύρια το χρόνο στο Μαλή η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας, της ε, αγροτικής υπαίθρου και με κατασκευή αεροδρόμων και δρόμων και η Αλγερία θα το θίξει σίγουρα το, στάνισή του Φθινοπόρου για την διασαχάρια οδό και άλλα για την ανάπτυξη, ε, μάλλον δεν πηγαίνει τίποτα για την ε, ασφάλεια. Ε, εντάξει, το κάνουμε για την ανάπτυξη, αλλά θα πρέπει να δούμε και τα δύο. Εδώ ομολογώ την άγνοια μου. Δεν ήξερα ότι υπάρχει μια εκμετάλλευση στο Μαλί ουρανίου. στο Νίγερα, ναι, αλλά δεν το κατάλαβα και πολύ καλά πάνω ναι, στον Νίγερα. Ε, διεξάγονται ιδιαίτερε έντερε συζητήσει γιατί γίνεται το πώ θα ωφεληθεί ο ντόπιο πληθυσμό από την εξόριξη του ουρανίου και θα πρέπει να το δούμε και πώ θα μπορούμε να βοηθήσουμε από πλάση Ευρωπαϊκή Ένωση για το θέμα αυτό. Ακόμα το άλλο θέμα που θίγετε εσεί, ναι, ήταν και το δυσκολότερο και μάλιστα για όλου μα. Να δούμε τι θα κάνουμε για την όλη οργάνωση ασφάλεια, πώ θα την ενισχύσουμε στι χώρε εκείνε που υπάρχει μια τάση για τι κυβερνήσει και μια διάθεση. Όλα αυτά να τα κάνει η κυβέρνηση για να επιτεθεί κατά τη ανταπολίτευση. Ε, η κυρία Άστον ε, διέκοψε, πάγωσε ένα πρόγραμμα για την Ιεμένη για την βελτίωση της οργάνωσης των προϊστορικών. Και αυτό για πολύ καλούς ε, λόγους, ε, γιατί βλέπουμε τι γίνεται τώρα στην σημερινή κατάσταση. Αυτό μας οδήγησε προς τα εκεί. Δεν είναι πάντα όμως ε, μαύρο-άσπρο το πράγμα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την προσέγγιση, τη δικαστική, την ποινική, την αστυνομική, να την βοηθήσουμε και για τις στρατιωτικές δυνάμεις που να έχουν ένα περισσότερο κλασικό ρόλο. Και ταυτόχρονα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ιδιαίτερα να επραγνυπνούμε για να μπορέσουν όλα αυτά να πάνε σε άλλους στόχους. Αυτά λοιπόν. Νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα να προσέχουμε το τι γίνεται. Απόλυτο δίκιο έχετε. Και για την Αίγυπτο τώρα. Όχι είναι η απάντηση. Από ό,τι γνωρίζω τουλάχιστον δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση του συστήματος ασφάλειας. Χρειάζονται τρόμερες ε, προσπάθειες και οι αρχές της Αιγύπτου δεν μας ζήτησαν τίποτα προς το παρόν. Αυτό το ίδιο και για την Τινησία. Νομίζω ότι έχει περισσότερη προτεραιότητα εκεί, υψηλότερη προτεραιότητα και υπάρχει στρατικό μηχανικό ισχυρό, αλλά θα πρέπει να δούμε και από δικαστική πλευρά μια κατάλληλη προσέγγιση. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν ένα από τους όλου παράγοντε τη εξίσωσης. Θα πρέπει να δούμε όσο μπορούμε να πιέσουμε χάρη στη χρηματοδοτησή μα ώστε αυτά τα κράτη να τα πείσουμε, να μα αφήσουν να του βοηθήσουμε. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ντεκερχόπ ε, για κύριε Ντεκέρχοφ για την ε, παρουσία και για αυτήν την ε, πλήρη σας παρουσίαση όλων αυτών των ζητημάτων. Ε, ελπίζω να σας ξαναδούμε σύντομα. Αν συμφωνείτε, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια και νομίζω ότι θα είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε επίσης, πέρα από τα ζητήματα που συζητήθηκαν και που είναι πολύ σημαντικά και δομικά, να παρακολουθήσουμε όλες τις πληροφορίες που μπορούν να προέλθουν από ε, την ε, κατάσταση που θα διαμορφωθεί μετά ε, το θάνατο του Οσάμα Μπιν Λάντεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ξαναβρεθούμε αύριο σε συνεργασία με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων για την συνεδρίαση με την Επίτροπο Γεωργίευα.